So, we continue... Λοιπόν, το σημείο 27. Ακρόαση για τις μετατροπές, διασπάσεις και την ψηφιοποίηση. Νέες δυνατότητες ε, για τις εταιρείες στην Ένωση. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή υπέβαλε το πακέτο για το εταιρικό δίκαιο, δύο νομοθετικές προτάσεις, στις 25 Απριλίου τρέχοντος για περισσότερη ελαστικότητα, επιτρέποντας διαμεθοριακές μετατροπές και διασπάσεις και τον εξυγχρονισμό μέσω της ψηφιοποίησης. Η Επιτροπή προσπάθησε να συνοδεύσει τα μέτρα αυτά με τις αναγκαίες εγγυήσεις. Η ακρόαση έχει τρία τμήματα. Κάθε ομιλητή θα έχει 7 λεπτά για την αρχική παρουσίαση. Μετά θα έχουμε συζήτηση θα πάρουν πρώτα το λόγο οι η κυρία Ρέγνερ και ο κύριος Γεύκα. Και αν κάποιοι από τους ομιλητές μας θέλουν να σχολιάσουν και άλλα θέματα του πακέτου, θα έχουν τη δυνατότητα. Λοιπόν, μεταξύ των διακεκριμένων ε, ομιλητών που έχουμε μαζί μας, πρώτα απ' όλα ο κύριος Βόλφκαν Κοβάλσκι από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση της Νομοσπονδίας σε αυτή τη τόσο σημαντική και πολύ χρήσιμη σε αυτή τη φάση ακρόαση αγαπητοί συνάδελφοι. Προέρχεστε από διάφορα κράτη-μέλη με διαφορετικές παραδόσεις και νοοτροπίες. Στις χώρες σας επιτρέπεται μια εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της, να μετατραπεί ή να διασπαστεί. Στις περισσότερες ε, χώρες αυτό δεν επιτρέπεται η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθούν εναρμονισμένοι ευρωπαϊκοί κανόνες όπως έχει κάνει και ασυγχωνεύσει στο παρελθόν αλλά αγνώρισε το γεγονός ότι στα κράτη-μέλη όπου δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί η έδρα ή να διασπαστεί μια εταιρεία ή να μετατραπεί γενικά δεν υπάρχουν βέβαια κανόνες για πληροφόρηση, διαβούλευση και συμμετοχή Οπότε, η πρόταση είναι πολύ μονόπλευρη και ιδιαίτερα φιλική προς τις επιχειρήσεις. Έχουμε γενικά κανόνες για την πληροφόρηση και την διαβούλευση. Δεν είναι ούτως ή άλλως πολύ ρωμαλές και για τα εργασιακά συμβούλια. Στα περισσότερα κράτη-μέλη έχουμε κανόνες ε, για την εκπροσώπηση σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου. Η καλύτερη προσέγγιση κατά τη γνώμη μας θα ήταν όπως και στο καταστατικό για τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες του 2001, να έχουμε μια διτή προσέγγιση. Να είναι ευκολότερο να μετακινηθούν οι εταιρείε και να δώσουμε και στους εργαζόμενους λόγο για αυτές τις ε, ενέργειες. Για παράδειγμα, να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στο, στα διοικητικά συμβούλια. Όμως δεν αξιοποίησε η Κομισιόν αυτή την ευκαιρία. Τώρα το Κοινοβούλιο πρέπει λοιπόν να διορθώσει την κατάσταση. Πρώτα απ' όλα για την ενιαία έδρα. Αυτό αποκλεί τις εταιρείε γραμματοκιβώτια και πρέπει να εδραιωθεί. Όπως ε, έχει εδραιωθεί στο νομοθέτημα για την Ευρωπαϊκή ε, Εταιρεία. Όμως η Κομισιόν λέει ότι δεν είναι δυνατή πλέον μια τέτοια προσέγγιση. Προτείνει μόνο κάποια κριτήρια δεν νομίζουμε ότι είναι ασφαλή. Μπορεί να υπάρξει τεράστια αύξηση των εταιριών γραμματοκιβωτίων αν μείνει όπως είναι το κείμενο. Και στην Ευρώπη έχουμε ήδη περίπου 500.000 τέτοιου τύπου εταιρείες. Σε μια δημοκρατία ο νομοθέτης μπορεί να τροποποιήσει τον νόμο. Υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Ξέρουμε λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βελτιώσει την πρόταση. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε περισσότερες τέτοιες εταιρείε πινακίδες που δεν πληρώνουν ε, για την κοινωνική ασφάλιση, που δεν φορολογούνται, που δεν υπόκειται σε κανένα εθνικό νόμο και που δεν διασφαλίζουν τα δικαιώματα ούτε των πιστωτών των εργαζομένων. Δεύτερο θέμα. Εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια. Εδώ και πολύ καιρό το Ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων έχει παρουσιάσει πολύ απλές, ευλίγιστες και ε, μη γραφειοκρατικές προτάσεις. Είναι το λεγόμενο σύστημα κυλιόμενη σκάλα. Προτείνει μία καινοτόμο συνεργασία μεταξύ των διαφόρων συστημάτων. Λέει ότι αν μια επιχείρηση έχει πάνω από 50 εργαζόμενους, δηλαδή πολύ μικρές επιχειρήσεις, εξαιρούνται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, θέλουμε δύο εκπροσώπους τα διοικητικά συμβούλια. Πάνω από 250 εργαζόμενοι, θέλουμε να υπάρχει ένα τρίτο. Και αν έχει πάνω από ε, χίλιου, θέλουμε τι μισέ έδρε. Η πρόταση αυτή είναι πολύ απλούστερη και μη γραφειοκρατική από του κανόνε αυτού. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε ένα φάκελο επάνω. Εάν διορθωθούν αυτά τα δύο κενά από το Κοινοβούλιο, όπως ελπίζουμε, η συνομοσπονδία μας ε, δεν θα αντιτίθετο πλέον. Αλλά σήμερα δεν θεωρούμε ότι είναι καν μισογεμάτο το ποτήρι. Μόνο κατά το 1 τρίτο θεωρούμε ότι είναι γεμάτο. Και κάτι άλλο. Έχουμε πολλές αμφιβολίες για την ανάγκη διάσπασης εταιριών. Θα σας παρακαλούσαμε να απορρίψετε αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχουν ε, πολλά κίνητρα σε αυτές τις προτάσεις για να παρακαμφθούν νόμοι και επειδή επίκυνται οι ευρωεκλογέ, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αυτή την πρόταση πολύ πιο ε, ρωμαλαία, πολύ πιο ασφαλή για τους εργαζόμενους. Η πρόταση πρέπει να μην είναι μια πρόταση όπου κερδίζουν οι εργοδότες και χάνουν οι εργαζόμενοι, πρέπει να είναι μια πρόταση όπου όλοι κερδίζουν. Αν δεν τροποποιηθεί, η πρόταση αυτή εξασφαλίζει ισότιμο ανταγωνισμό για τους εργοδότες, αλλά αδικεί τους εργαζόμενους. Δεν μπορεί να είναι δίκαιο κάτι τέτοιο. Αλλά για να μην παρεξηγηθώ, δεν θέλουμε να απορρίψουμε τις προτάσεις. Θέλουμε να τις βελτιώσουμε. Θα θέλαμε εσείς να βελτιώσετε το κείμενο. Θέλουμε αυτή τη στιγμή να υπάρξει περισσότερη δημοκρατία στον τόπο εργασία. Κάνουμε μια εκστρατεία προς αυτή την κατεύθυνση και έχουμε εκπονήσει μια ευρωπαϊκή έκκληση για περισσότερη συμμετοχή των ε, εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Έχουμε ήδη 600 υπογραφές από πανεπιστημιακούς ε, και ευρωβουλευτές και 45 γενικούς γραμματείς νομοσπονδιών ε, εργαζομένων από 42 χώρες. Θα θέλαμε αυτό το σαφές αίτημα να το λάβετε υπόψη. Η Επιτροπή μας για το Εταιρικό Δίκαιο συνεδρίασε χθες και σας παρουσιάζω τώρα την ε, ομόφωνη άποψη αυτής της Επιτροπής που είναι ε, ένα πολύ σημαντικό σώμα ενώ το ανώτερο σώμα μας θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Σόφια όπου θα μπορείτε να δείτε μετά στο site μας την τελειωτική μας άποψη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα Πέδρο Ολιβέρα, διευθυντή ε, Νομικών Θεμάτων του οργανισμού Business Europe. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Κοινοβουλίου θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση εκ μέρους της Business Europe, η οποία εκπροσωπεί εταιρεία σε 34 διαφορετικές χώρες. Αυτό το πακέτο προτάσεων για το εταιρικό δίκαιο είναι πολύ ουσιαστικό θέμα για τις επιχειρήσεις. Είναι ουσιαστικό στοιχείο του εμπορικού δικαίου και είναι κάτι που το ζητούσαμε εδώ και πολύ καιρό. Ξεκινώ λοιπόν ε, με θετικό πνεύμα, καλωσορίζοντας την πρόταση. Και στο δελτίο τύπου που εκδώσαμε όταν δημοσιοποιήθηκε η πρόταση η νομοθετική τον Απρίλιο, το την καλωσορίσαμε για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα για λόγους αρχής, ε, γιατί επί 30 χρόνια ζητούσαμε να γίνει ε, θεσμοθετηθεί η ελευθερία σύστασης επιχειρήσεων και επίσης ζητούσαμε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τις μεταβολές και τις διασπάσεις, οι οποίες δημιουργούσαν εμπόδια σε αυτή την ελευθερία. Και βεβαίως είχαν υπάρξει εξελίξεις, είχαμε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αν και αυτές οι εξελίξεις ήταν θετικές, δεν αρκούσαν τα δικαστήρια, έχουν τα όρια τους. Χρειάζονται ουσιαστικοί κανόνες για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου. Ο δεύτερος λόγος, τον οποίο καλωσορίσαμε την πρόταση, ήταν η ψηφιοποίηση η χρήση της πληροφορικής είναι ένα τρένο που δεν πρέπει να χάσουμε, θα πρέπει και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπουν στον 21ο αιώνα. Όπως θα διαπιστώσει κανείς από την πρώτη ανάγνωση της πρότασης, είναι περίπλοκη, είναι τεχνική, χρειάστηκε χρόνος. Γι' αυτόν τον λόγο επίσης και η Business Europe δεν έχει καταλήξει ακόμα στην θέση της, στην τελική, την οποία θα οριστικοποιήσουμε στις επόμενες εβδομάδες. Επομένως, η παρουσίαση μου σήμερα είναι μια πρώτη αξιολόγηση της πρότασης. Και αργότερα θα μοιραστούμε και τις υπόλοιπες μας απόψεις για το θέμα. Εγώ θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο ζήτημα της κινητικότητας, αυτό το σκέλος της πρότασης, Και τρεις είναι οι βασικές ιδέες που θα προσπαθήσω να παρουσιάσω σήμερα για το θέμα αυτό, που μπορώ να τις περιγράψω και με τρία, τρεις λέξεις. Την διευκόλυνση, την περιπλοκότητα και τις ασφαλιστικές δικλείδες. Τι εννοώ με την ε, διευκόλυνση. Δείτε το ζήτημα από την πλευρά των επιχειρήσεων. Χρειάζεται, ε, χρειαζόμαστε ε, πάρα πολύ να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση της επιχείρησης, γιατί τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν έρθει πολλές νομικές, νομοθετικές πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές από αυτές τις έχει υποστηρίξει και παρακολουθήσει και η Επιτροπή σε Είναι τα ζητήματα της γεωγραφικής προέλευσης, της προστασίας του καταναλωτή και άλλα πολλά. Τι εννοώ λοιπόν με τη διευκόλυνση. Εννοώ κανόνες και ε, πλαίσια τα οποία θα μπορέσουν να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και θα δημιουργήσουν ένα υγιές πλαίσιο για αυτήν. Σε όλη τη διάρκεια ζωής μιας επιχείρησης, από την σύσταση της, κατά τη διάρκεια της άσκησης της διοίκησης σε αυτήν, την πρόσβαση σε κεφάλαια και επίσης όταν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει κανείς τις πρώτες δυσκολίες. Αυτό το πακέτο λοιπόν για το εταιρικό δίκαιο είναι μια μορφή διευκόλυνση προς τις επιχειρήσεις κατά την άποψή μας. Είναι μια πολύ σημαντική πρόταση και ελπίζουμε να βρεθεί ε, μια ισορροπημένη λύση. Το δεύτερο θέμα είναι η πολυπλοκότητα. Μας ικανοποιούν οι διαδικασίες που προβλέπονται, όμως υπάρχουν κάποια στοιχεία της πρότασης που αναρωτιόμαστε πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη. Έχω προετοιμάσει και μια μικρή διαφάνεια για να σας δείξω με οπτικό τρόπο ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για τις ε, μεταβολές και με τις διασπάσεις είναι κάπως παρόμοια τα πράγματα οι συγχωνεύσει είναι λιγότερο περίπλοκε, αλλά νομίζω ακόμα και βλέποντα την διαφάνεια καταλαβαίνετε την πολυπλοκότητα του συστήματο. Για να κάνει κανεί μια μεταβολή, σύμφωνα με το, την πρόταση, για να ολοκληρώσει κανεί όλα τα στάδια, δεν του αρκεί ένα δικηγόρος, χρειάζεται έναν άνθρωπο που να γνωρίζει κβαντική φυσική. Με λίγα λόγια σας λέω ότι οι διαδικασίες που προβλέπονται είναι πολύ περίπλοκες, είναι ε, κοστοβόρες, θα κοστίζουν πολύ και επίσης θα υπάρχει και ε, θα υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις. για τέτοιου τύπου μεταβολές στις εταιρείε, στις επιχειρήσεις, θα έπρεπε να έχουμε διαδικασίες πολύ απλούστερες και εύκολες. Το τρίτο μήνυμα θα ήθελα να σας ε, στείλω σήμερα έχει σχέση με τις ασφαλιστικές δικλείδες. Οι επιχειρήσεις δεν δημιουργούνται για να κάνουν απάτες. Στόχος των επιχειρήσεων είναι να παράγουν αξία, προστιθέμενη αξία, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να προχωρήσει η οικονομία. Ε, βεβαίως υπάρχει κίνδυνος της απάτης, υπάρχουν κάποια σάπια Μίλα, αλλά αυτό δεν είναι ο κανόνας. Στην εξαίρεση. Επομένως, όπως πάντοτε στο εταιρικό δίκαιο, χρειάζεται να έχουμε και κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες για τη σύσταση, για την δυνατότητά της να μεταβάλει την έδρα της, για τη μεταβολή της μετοχικής της σύνθεσης, σε περιπτώσεις διάλυσης ή χρεοκοπίας. Ε, Βεβαίω χρειάζονται ασφαλιστικέ δικλείδε για όλα αυτά. Κανεί δεν τον αμφισβητεί. Για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων. Είτε πρόκειται για πιστωτέ, που είναι με τη σειρά του ε, ε, ε, και, αυτές και αυτέ τι επιχειρήσει ή άλλε εταιρείε, ε, και φυσικά του εργαζόμενου, όπω επίση και του πελάτε του κράτου. Πιστεύουμε όμως ότι η πρόταση της Επιτροπής το παρακάνει. Με ε, όλες αυτές τις απαιτήσεις που εισάγει, τις οποίες θεωρούμε μη αναλογικές, και πιστεύουμε ότι προέρχονται από μια αρνητική αντίληψη για την επιχειρηματικότητα αναφέρονται όροι όπως για παράδειγμα ε, διευθετήσεις με σκοπό την ε, φοροαποφυγή κτλ. Μιλούμε εδώ για διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται σε κάθε μια από τα στάδια της, τους κύκλου ζωής μιας επιχείρησης. Δεν είναι λογικό να θεωρείται η επιχείρηση, η εταιρεία καταρχήν ένοχη. όταν πληρεί κάποια κριτήρια, όταν δεν ε, υπάρχει καμία ένδειξη ότι κάτι πάει στραβά, ε, θα πρέπει η διαδικασία να είναι απλή. Δεν μπορούμε να ξεκινούμε θεωρώντας ότι πρέπει να αποδείξει την αθότητά της. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει μια ε, να, να υπάρχει μια δυνατότητα να μπορούν τα κράτη-μέλη να κάνουν μια αξιολόγηση σε δεύτερο επίπεδο, βαθύτερη, μόνο όταν έχουν υπάρξει κάποιες ενδείξεις, όταν για παράδειγμα έχουν υποβληθεί κάποιες καταγγελίες από μετόχους, αλλά όχι αυτό να γίνεται σε κάθε περίπτωση. Επίση, οι επιχειρήσει που εκπροσωπούμε δεν είναι ικανοποιημένε από τις προβλέψεις σε αυτή την πρόταση σε σχέση με τους εργαζόμενους εάν ε, δείτε τις μελέτες που έγιναν πριν από την οδηγία για τις συγχωνεύσεις. Ένα από τα συμπεράσματα ήταν ότι αυτές οι διατάξεις έκαναν τη λειτουργία των επιχειρήσεων πιο περίπλοκη και αυτό έχει αποτρέψει τις επιχειρήσεις να επιλέξουν κάποιες από τις δυνατότητες που τους έδινε η πρόταση. Πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν οι όποιες διατάξεις να είναι απλές, εξασφαλίζοντας βέβαια αυτό που πρέπει να εξασφαλιστεί. Όμως εμείς αυτό που βλέπουμε ότι προστίθονται και άλλες προϋποθέσεις και μάλιστα ίσως εισάγονται και κάποιες επικαλύψεις ε, με υφιστάμενη νομοθεσία. Κατά την άποψή μας λοιπόν, αξιότιμο μέλη του Κοινοβουλίου, πρέπει να εργαστούμε περισσότερο για το θέμα, να το αναλύσουμε περισσότερο. Η Business Europe από την πλευρά της θα το πράξει, θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια επικοδομητική στάση, όπως έλεγε ο συνάδελφο μου πριν. Ε, όμως θα ε, σας επισημάνουμε τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει αυτή η πρόταση, γιατί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση μια τέτοια πρόταση να αυξήσει το κόστος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Αυτό ήταν το πρώτο τμήμα που ονομάσαμε η άποψη των κοινωνικών εταίρων. να πάμε στο δεύτερο, να ρωτήσω την κυρία Ρέγκνερ, ο συζηγήτρια, αν έχει ερωτήσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις σας. Από τη σκοπιά δηλαδή των κοινωνικών εταίρων. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σας θέσω. Αντίστροφα που θα έλεγα ρωτάω ερωτήσεις που συνήθως απευθύνονται στο Business Europe από τα συνδικάτα. Οπότε ως εκπρόσωπος του Business Europe να πω το εξή. Αναφέρθηκε από τον συνάδελφο από τα συνδικάτα ότι υπάρχουν γύρω στις 500.000 εταιρείε γραμματοκιβώτια. Αυτό θα θέλαμε να το αποφύγουμε, γιατί δεν είμαι εγώ μόνο μέλος εδώ σε αυτή την επιτροπή, αλλά ασχολήθηκα και με τα Panama Papers, τα Paradise Papers και ένα ολόκληρο φάσμα αρνητικού αντικτύπου που εξετάσαμε. Οπότε όταν λέμε ότι χρειαζόμαστε διευκολύνσεις και ότι τα πράγματα πάνε πολύ μακριά, εσείς τι θα προτείνατε ώστε να μειώσουμε αυτόν τον αριθμό των εταιριών γραμματοκιβώτια. Είδαμε ότι έχουμε κανόνες εταιρικού δικαίου, όμως έχουμε συστήματα που ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Οπότε κατά κάποιο τρόπο η μεγάλη μας πρόκληση είναι να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Να έχουμε δηλαδή ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο, αφενός και αφετέρου να έχουμε εθνικές αρχές οι οποίες ελέγχουν τους επιμέρους κανόνες τους εθνικούς. Πρώτη ρώτηση αυτή. Δεύτερη, αναφερθήκατε στους διευκολυντές, τους enablers. Μήπως θα ήταν καλύτερο για σας να έχουμε μια πρόταση που βεβαίως δεν έχετε τώρα, αλλά τέλος πάντων για τη μεταφορά της έδρας, όπως λέμε στα γερμανικά. Δηλαδή το εργαλείο που αφορά τις προτάσεις μετατροπές, ηχονεύσεις, διασπάσεις. Μήπως θα ήταν τότε πιο εύκολο να έχουμε τη μεταφορά της έδρας από το να λέτε εσείς ότι ε, υπάρχει αυτή τη στιγμή και συζητείτε. Και άλλη μια ερώτηση προς τον κύριο Κοβάλσκι. Μήπως υπάρχει μια αντίφαση. Έχουμε τις τέσσερις βασικές ελευθερίες. Αφενός και αφετέρου έχουμε πάντοτε τα παραθυράκια και τις δράσεις κατά των εργαζομένων. Οπότε εσείς τι προτείνετε. Εντάξει, μιλήσατε για, εταιρείε ε, γραμματοκιβώτια και τις αρνητικές επιπτώσεις αλλά κατά την άποψή σας ξεκάθαρα ποιο θα ήταν το κατάλληλο μέτρο για να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη κατάσταση γιατί αυτό το αντιμετωπίζουμε συνεχώς βλέπουμε ότι προβλήματα υπάρχουν Ωραία, αλλά ποιο θα ήταν ένα έτσι ισχυρό εργαλείο καταπολέμησης που θα ενισχύσει αυτές τις δικλείδες που υπάρχουν. Τι προτείνετε εσείς λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Κιτάντ. Ήθελα και αυτή να θέσει ένα ερώτημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες εισηγήσει σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι και τους δυο σας, αλλά και την Κομισιόν. Η Κομισιόν ίσως στη συνέχεια να απαντήσει ένα κύριο στοιχείο αυτής της διαδικασίας για μετατροπές συγχωνεύσεις διασπάσεις είναι το να αποτρέψουμε τις μετατροπές όταν ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει κατάχρηση ή υπάρχουν ε, τεχνητές ρυθμίσεις για να αποκομίσει κανείς φορολογικό πλεονέκτημα ή αν υπάρχουν ε, δικαιώματα των μελών τη μειοψηφίας τα οποία πλήττονται. Αυτό αναφέρεται συγκεκριμένα στο 86 γ3 της πρότασης. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς ακριβώς ορίζεται το φορολογικό πλεονέκτημα το οποίο είναι αθέμητο. Αθέμητο φορολογικό πλεονέκτημα. Πώς το ορίζεται και ποιες είναι οι μακροχρόνιες επιπτώσεις αυτού του σκεπτικού. Δηλαδή, όταν θέλουμε να αποτρέψουμε τις δομές των εταιριών ε, γραμματοκιβώτια οι οποίες παραβιάζουν εθνικούς, ε, εθνικούς νόμους. Ε, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ναι, μήπως θα θέλατε να απαντήσετε σύντομα. Ναι, πολύ σύντομα για τις διάφορες ερωτήσεις. 500.000 εταιρείε γραμματοκιβώτια. Αυτός ο αριθμός δεν ξέρω από πού προκύπτει και θα ήταν καλό να μάθουμε από πού βγήκαν αυτές οι στατιστικές και με ποια μεθοδολογία. Αυτές οι εταιρείε είναι εταιρείε ε, κέλυφος ή έχουν κάποια εταιρική τέλο πάντων δραστηριότητα, αυτό θα πρέπει να το ελέγξουμε. Τώρα, αυτό που θα θέλαμε να μειώσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι οι καταχρήσεις. Και οι εταιρείε γραμματοκιβώτιο όντως είναι ένας τρόπος από αυτούς που χρησιμοποιούνται για τις καταχρήσεις αυτές. Δεν θεωρούμε ότι το εταιρικό δίκαιο αποτελεί πανάκια. Έχουμε και άλλους τομείς του νόμου, φορολογική νομοθεσία, έχουμε την οδηγία για την φόρα αποφυγή που υιοθετήθηκε πέρσι και πρόκειται να εφαρμοστεί και εκεί έχουμε πολλές διατάξεις που αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από το να καταχρούνται του συστήματος. Επίσης, αν θέλουμε να λύσουμε το θέμα των εργαζομένων και του εργατικού δικαίου, ίσως το εταιρικό δίκαιο να μην είναι το καταλληλότερο μέρος για να γίνει αυτό. Έχουμε το κοινωνικό διάλογο, έχουμε διατάξεις από τη συνθήκη που κάνουν προβλέψεις. Οπότε, για να απαντήσω στο πρώτο ερώτημά σας, δεν νομίζω ότι το εταιρικό δίκαιο αποτελεί πούμε, το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα λύσουμε όλα τα προβλήματα που έχουμε στην Ένωση. Μετά, για τι διαφορέ που η κυρία Ρέκνερ σωστά ανέφερε, όντω υπάρχουν πολλέ διαφορέ όσον αφορά του κανόνε τη χώρε μέλη. Ακόμα και για τη σύσταση των επιχειρήσεων, τι έδρε, τι πραγματικέ έδρε κλπ. Έχουμε και την οδηγία για τι συγχωνεύσει. πολύ επιτυχή. Είχαμε 200% αύξηση μετά την εφαρμογή της. Έχουμε λοιπόν κάποια εναρμόνιση που σε σχέση με το εταιρικό δίκαιο είναι αποτελεσματική. Ελπίζουμε ότι λόγω αυτού του γεγονότο θα μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι το οποίο θα αποδειχτεί χρήσιμο. Αναφερθήκατε στη μεταφορά τη έδρα, κατά πόσο αυτό αρκεί. Όχι, δεν αρκεί, επειδή καλύπτει μόνο ένα τμήμα των λειτουργιών της επιχείρησης. Θα θέλαμε να έχουμε κάτι το οποίο να είναι πιο περιεκτικό. Και νομίζω έχει έρθει η ώρα να το κάνουμε. Η κυρία Γιούταλα μίλησε για τα κριτήρια για αυτή την έκφραση artificial arrangement τεχνητές διαδικασίες δεν ξέρουμε τώρα κατά πόσο υπάρχει αντίκρισμα αυτής της έκφρασης στη νέα νομοθεσία. Δεν ξέρουμε κατά πόσο εδώ έχουμε ας πούμε νέες διατάξεις που αφορούν καταστάσεις όπου έχουμε καταχρήσεις ευρείες. Εδώ αυτό δεν καλύπτεται. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε και εμείς ακριβώς πώς αυτή η έκφραση θα προσδιοριστεί ή θα οριστεί σε συγκεκριμένο επίπεδο. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι επιχειρήσεις καταρχάς ακολουθούν την αρχή ότι μπορούν να μετακινηθούν στην Ένωση ακριβώς για να επωφεληθούν καλύτερων φορολογικών διατάξεων. Τώρα, όταν καταχράσει αυτό το γεγονότο, κάτι δεν πάει καλά, λέει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου ότι βεβαίω μπορεί να μετακινηθεί στα θέση να έχει καλύτερη φορολόγηση. Δεν νομίζω λοιπόν ότι όλες οι μετακινήσεις είναι λάθος. Μπορούν να μετακινηθούν επιχειρήσεις συμμεριζόμαστε το ενδιαφέρον που δείχνετε για να το προσδιορίσουμε αυτό και να είναι σωστό. Τελικά όμως να μην ξεχνάμε και τις βασικές αρχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σύντομη απάντηση από εσά, παρακαλώ. Δεν θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω. Νομίζω είναι πολύ εύκολο να υπερχαράξουμε το θέμα των επιχειρήσεων στο, ε, στο εργατικό δίκαιο. Εδώ στις εταιρείε έχουμε όλες αυτές τις πλευρές. Έχουμε τους εργοδότες, έχουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, έχουμε τους εργαζόμενους, οπότε δεν γίνεται μόνο να κάνουμε κάτι αποσπασματικά μόνο για τους εργαζόμενους ή μόνο για το λειτουργικό κομμάτι της επιχείρησης. Αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της επιχείρησης οι εργαζόμενοι. Τώρα για αυτές τις τεχνητές διαδικασίες Ναι, για τις συγχωνεύσεις μιλάμε, αλλά δεν θα πέρασω αυτό στη συνέχεια. 90% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι επιχειρήσεις κέλυφος και Και έχουμε τώρα αυτή την οδηγία εδώ και δύο δεκαετίες όπου οι επιχειρήσει όπου όντω συμμετέχουν εργαζόμενοι γύρω στα 150. Δεν μπορείτε να το θεωρήσετε αυτό success story. Δεν μπορώ να σα πω γιατί, εντάξει είναι η στιγμή. Τώρα για τι συγχωνεύσει. Λέει η Κομισιόν ότι αυξήθηκαν οι συνεργειακέ ε, συγχωνεύσει κατά 173%. Ε, Όπω είπε η ίδια αυτό Αλλά εξαρτάται από ποια χρονιά κοιτάτε. Αν κοιτάξουμε την περίοδο 2008-2015, η αύξηση ήταν μόνο 30%. Και το σύνολο, γιατί ξέρετε ότι έχουμε 22 εκατομμύρια επιχειρήσεις στην Ευρώπη, πόσες χρησιμοποίησαν αυτή τη δυνατότητα μεταξύ 200 και 300 ετησίως. Μην υπερβάλλετε λοιπόν. Αυτές οι τεχνητές διαδικασίες ε, είναι πολλές Μισό εκατομμύριο σχέση με 22 εκατομμύρια είναι πολύ μεγάλος αριθμός, οπότε θα πρέπει εμείς να διασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι περισσότερες. Τώρα, για το αν έχω μια ξεκάθαρη πρόταση για το πώς θα είναι στεγανή η διαδικασία για την ψηφιοποίηση, τι να σας πω. Νομίζω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, διευθυντές, ιδιοκτήτες κτλ. θα πρέπει να ελέγχονται διαδικαστικά σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες. Εκεί θα υπάρξουν προτάσεις, αλλά αυτές οι τεχνητές διαδικασίες δεν είναι αυτό που επιθυμούμε. Δεν θέλουμε οι επιχειρήσεις κυρίως να ασχολούνται με την αποφυγή της φορολογίας και τη μείωσή της. Νομίζω ότι μια επιχείρηση σαν την Polbot στην Πολωνία η οποία μετέφερε την έδρα της απλά και μόνο για να μειώσει τη φορολογία της χωρίς ακριβώς να μεταφέρει καμία εταιρική δραστηριότητα γίνεται είναι θεμητό, επιτρεπτό το θέλουμε όμως αυτό γιατί λέει η αξιολόγηση αντικτύπου ότι θα υπάρχει χαμηλότερη φορολογική συμβολή σε κάποιες χώρες μέλη. Το θέλουμε αυτό. Οπότε θα έχουμε χαμηλότερη κοινωνική πρόνοια από τις εισφορές αυτής της εταιρεία. Αυτό θέλουμε. Υπάρχουν λοιπόν πολλές δυνατότητες παράκαμψης και θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε βέβαια όλα αυτά όταν κάνουμε στεγανό το πακέτο για την ψηφιοποίηση και για τις ε, μετατροπές ε, βεβαίως θα πρέπει να συζητήσουμε και με το εργατικό δυναμικό να συζητήσουμε και με άλλους. Αν έχετε ένα καλό εταιρικό σχέδιο και αν θέλετε να μετακινηθείτε για θεμητούς λόγους, τότε το εργατικό, εργατικό δυναμικό μπορεί να μην αντιταχθεί. Και είναι πάντοτε χρήσιμο να συζητά κανείς με τους ε, εμπλεκόμενους και νομίζω ότι το ίδιο θα κάνουμε σε αυτό το πλαίσιο της οδηγίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που επιμένω για συντομία γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει. Αλλά να θέσω μια ερώτηση στον κύριο Κοβάλσκι. Σε μία πρόταση παρακαλώ. Από πού αντλείτε τα στοιχεία σας. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Και θα σας πω. Ωραία, μπορείτε να απαντήσετε μετά τις επόμενες ομιλίες. Έτσι έχετε όλο το χρόνο που χρειάζεστε για να ψάξετε για μία απάντηση. Πάμε τώρα στο δεύτερο τμήμα της ακρόασης. Κίνδυνοι και ευκαιρίες. Να δώσω το λόγο στην κυρία Page Morrow, που είναι λέκτορας για την εταιρική διακυβέρνηση στο Πανεπιστήμιο του Κέντ. 7 λεπτά παρακαλώ κυρία μου. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας ενημερώσω για το πακέτο, για το εταιρικό δίκαιο, επειδή είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Θα επιχειρήσω να είμαι σύντομη γιατί λέτε ότι θέλει αυτή η νομοθεσία να βοηθήσει τις διαμεθοριακές επιχειρήσεις αλλά παράλληλα να βοηθήσει τους εργαζόμενους και να αποφύγει την ε, φόρο διαφυγή. Έχω εργαστεί για αυτούς τους τομείς. Υποθέτω ότι όλοι καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πακέτο. Οπότε θα ασχοληθώ με πολύ συγκεκριμένα θέματα, όπου το Κοινοβούλιο μπορεί να επιφέρει ίσως και βελτιώσεις. Μετά ο καθηγητής ο κ. Κόνακ θα σας πει περισσότερα. Με συγχωρείτε, έχω το κουμπί αυτό που λέει να ε, μιλάτε αργά. Ακόμη και όταν μιλάει πολύ αργά ο μιλητής. Α, ωραία, βλέπω διορθώθηκε. Ευχαριστώ. Για την οδηγία, για τις διαμεθοριακές ε, μετατροπές, συγχωνεύσεις και διαιρέσεις, διασπάσεις μάλλον. Ο νόμος που προστατεύει την ελεύθερη κυκλοφορία έχει επιτρέψει ιδιαίτερα και ενθαρρύνει τις εταιρείες πινακίδες. Αλλά έχει γίνει κατανοητή η κατάσταση αυτή και γίνεται προσπάθεια περιορισμού της, της για παράδειγμα μέσω της οδηγίας για τους ε, αποσπασμένους. Προβλέπεται τώρα ότι το κράτος προέλευσης μπορεί να περιορίσει αυτό το αυτή τη δυνατότητα αν υπάρχει δημόσιο συμφέρον. Το δικαστήριο και η νομολογία του λέει σαφώς ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να εγκρίνουν νομοθεσία για να αποφεύγεται η παράκαμψη της εθνικής νομοθεσίας. Η οδηγία αυτή προσπαθεί να διευκολύνει τις διαμεθοριακές επιχειρήσεις αλλά να παράλληλα να προστατεύσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Άρα δεν θέλουμε να αλλάξουμε τα συστήματα εθνικής φορολογίας, να μειώσουμε τους συντελεστές ή να περιορίσουμε την υποχρεωτική συμμετοχή των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια που είναι ε, υποχρεωτική με βάση την εταιρική διακυβέρνηση πολλά κράτη-μέλη. Το πακέτο αυτό στοχεύει να διευκολύνει τη δημιουργία σύστασης εταιριών που σημαίνει ε, γνήσια οικονομική δραστηριότητα στο κράτος ε, στο οποίο μεταφέρεται μια εταιρεία όπου δεν υπάρχει καμία ουσιώδη οικονομική δραστηριότητα ή αν θέλουν να αποφύγουν τη φορολογία και την εκπροσώπηση των εργαζομένων, τα κράτη-μέλη μπορούν να θεωρήσουν ότι αυτή η αναδιάρθρωση είναι τεχνητή, τεχνητό εγχείρημα και να τον μπλοκάρουν. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 7. Γενικά, το εταιρικό δίκαιο αυξάνει την βασική αρχή ε, του εταιρικού δικαίου στην Ευρώπη που είναι η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Υπάρχουν εξαιρέσει, όπως οι ιδεολογικές σκέψεις της ε, οδηγία για τους μετόχους. Αυτό δεν ε, μεταφέρεται σωστά στον δευτερογενή νόμο και πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει. Μια συγκεκριμένη πρόταση θα ήταν να μπει μια ρήτρα για τους εμπλεκομένους φορεί στο άρθρο 1 που θα λέει ότι τα διοικητικά συμβούλια είναι αρμόδια για την δίκηση τη εταιρεία προ το συμφέρον τη εταιρεία. Λαμβάνοντα υπόψη τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων και άλλων ε, συμμετεχόντων. Για να δημιουργηθεί ουσιώδη αξία. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της πρότασης είναι ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν μια διαδικασία για τις διαμεθοριακές μετατροπές και διασπάσεις οι Εθνικέ αρχές θα πρέπει να εξετάσουν τα έγγραφα των εταιριών και να δώσουν ένα ε, προκαταρκτικό πιστοποιητικό. Οι αρμόδιε αρχές του κράτους προέλευση θα εκδώσει αυτό το πιστοποιητικό αφού εξετάσει και εφόσον καταλήξει ότι αυτή η μετατροπή ή διάσπαση είναι νομότυπη και δεν θα επιτρέπεται καμία τέτοια δραστηριότητα, καμία τέτοια επιχείρηση, αν στόχος είναι άδικα φορολογικά πλεονεκτήματα ή ο περιορισμός των νομίμων δικαιωμάτων ε, των μετόχων ή των εργαζομένων ή των πιστωτών. Εάν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι υπάρχουν τέτοιες ε, προσπάθειες τεχνητής, τεχνητού εγχειρήματος, τότε μπορεί να λάβει μέτρα το κράτος προέλευσης, το αρχικό κράτος. Οι κανόνες όμως αυτή τη στιγμή δεν ισχύουν για τις διαμεθοριακές συγχωνεύσεις. Η πρόταση της Επιτροπής δεν το περιέχει. Αυτό δημιουργεί στην ουσία κέντρο ε, οι συγχωνεύσεις να οδηγήσουν σε αναδιαρθρώσεις που μετά κατόπιν θα μετατραπούν σε μετατροπές και διασπάσεις. Άρα η Επιτροπή σας θα μπορούσε ενδεχομένω να εξετάσει την τροπολόγηση του κειμένου ούτω ώστε αυτά τα τεχνητά εγχειρήματα να αφορούν και τι ε, διαμεθοριακέ συγχωνεύσει. Έτσι θα έχουμε ένα απόλυτα εναρμονισμένο σύστημα για διαμεθοριακέ αναδιαρθρώσει. Κάτι άλλο, σχετικό. Για να μην υπάρχουν κενά στην προστασία των άλλων ε, συμμετεχόντων, θα πρέπει να σεβόμεθα την αρχή του, της απαρίθμησης. Δηλαδή, μόνο οι ενέργειες που συγκεκριμένα επιτρέπονται από την οδηγία θα μπορούν να εκτελεστούν. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρξει ένα νέο άρθρο στην αρχή της οδηγίας που να διευκρινίζει οι μορφές αναδιάρθρωσης που αναφέρονται είναι οι μόνες μορφές που επιτρέπονται. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει εκ των υστέρων παρακολούθηση της εφαρμογής. Όλοι οι τεχνητοί διακανονισμοί τελικά μπορεί να γίνουν ε, σαφείς μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης. Έχουν γίνει διάφορες προτάσεις. Ποιος θα κάνει αυτούς τους ελέγχους, η Επιτροπή, το αρχικό κράτος, ή η προτινόμενη τώρα Ευρωπαϊκή ε, Εργασιακή Αρχή. Εντάξει, μπορεί να συζητηθεί, αλλά είναι σημαντικό θέμα. Πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω. Για την ψηφιοποίηση. Τα εξής. Οι Eurojust και άλλοι δήμονες έχουν εκφράσει ανησυχίες για ε, την πλήρη ψηφιοποίηση. Αυτό μπορεί να ευνοήσει την τρομοκρατία, το ξέπλυμα χρήματος, τη φοροαποφυγή και άλλες μορφές εγκληματικότητας. Μια απλή λύση θα ήταν να περιοριστεί η χρήση αυτής της επιγραμμικής διαδικασίας σε φυσικά πρόσωπα. Όχι νομικά. Δεύτερον, η επαλήθευση των στοιχείων των διευθυντών με βάση αυτή την πρόταση επαφείται στην εθνική νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση. Να υπάρχουν διασυνδεδεμένα μητρώα επιχειρήσεων. Και υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά την ποιότητα αυτών των ε, μητρώων. Πρέπει και αυτά να εξεταστούν. Τέλος. Χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια και εύκολη πρόσβαση του κοινού στα στοιχεία για την λειτουργία των εταιριών, τα οικονομικά στοιχεία. Η διασύνδεση, για παράδειγμα, της διασύνδεσης των, ε, εταιρικών μητρών θα βοηθούσε την ε, διαφάνεια αυτής της πληροφόρησης. Τα λέει αυτά η νέα οδηγία κατά του ξεπλήματος. Έτσι θα ήταν πολύ σαφέστερο ποιος είναι πίσω από κάθε εταιρεία. Λόγω του περιορισμένου χρόνου κλείνω στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο στον καθηγητή Κονάκ, καθηγητή εμπορικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να σας δώσω την, μια αξιολόγηση της πρότασης αυτής για το εταιρικό δίκαιο και όπως και οι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω από το ζήτημα της ψηφιοποίησης και μετά θα μιλήσουμε για τις μεταβολές. Αυτές οι δύο προτάσεις είναι κάτι που οι δεμπλεκόμενοι μέρη ενδιαφερόμενοι ζητούν εδώ και πολλά χρόνια. Με στόχο να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις ε, στην πρόσβασή τους στην ενιαία αγορά, να μπορούν να μεταβάλουν την έδρα τους και αυτό το ζητούν εδώ και 30 χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να συγχαρούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είχε το θάρρος να προχωρήσει στο θέμα αυτό. Γνωρίζουμε ότι με βάση την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη επιτρέπονται κάποια από αυτά τα πράγματα, αλλά ε, τώρα κωδικοποιούνται ε, έτσι ώστε να υπάρχει προστασία για όλους. Και αυτό είναι μια τεράστια ε, βελτίωση γιατί δημιουργεί ε, ασφάλεια δικαίου σε όλες τις περιπτώσεις. Αν δείτε τις δημόσιες διαβουλεύσεις που έχουν γίνει εδώ και 30 χρόνια, υπήρχε καθολική υποστήριξη των προτάσεων αυτών. Θεωρώ ότι και η πρωτοβουλία ψηφιοποίηση είναι ένα βήμα θετικό. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που έχουν ήδη ψηφιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τα μητρώα τους από το 2014 είχε γίνει μια προσπάθεια με την πρόταση για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία και βλέπω ότι στη νέα πρόταση της Επιτροπής έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παρατηρήσεις που είχαν υποβληθεί τότε. Για παράδειγμα για τα ζητήματα της καταπολέμησης του ξεπλήματος μαύρου ε, χρήματος, ε, της απάτης. Πιστεύω ότι η σύνταξη λοιπόν αυτής της πρότασης από την πλευρά της Επιτροπής έγινε λαμβάνοντας υπόψη ε, τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων και των απόψεων της ε, Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ε, και των συμβολεογράφων, δεν θέλω να μιλήσω εξ τους, αλλά διαπιστώνω ότι αυτή τη στιγμή την υποστηρίζουν την πρόταση. Θα βελτιωθεί η πρόσβαση λοιπόν στην ενιαία αγορά για όλες τις επιχειρήσεις και για τα παραρτήματά τους. Αυτός γενική αξιολόγηση. Ας δούμε λοιπόν τώρα το ζήτημα των μεταβολών διασπάσεων και συγχωνεύσεων διασυνοριακά. Και πάλι, αυτή η πρόταση οδηγίας έχει λάβει υπόψη της τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων. Το έκανε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδιαίτερα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θεωρώ ότι η, πρόταση, η προτινόμενη οδηγία δεν θα μειώσει την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ε, βεβαίως το εταιρικό δίκαιο δεν είναι εργατικό δίκαιο. Τα εργατικά θέματα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο εργατικό δίκαιο, αλλά έχουμε και άλλου που πρέπει να φροντίσουμε. Τα συμφέροντα του κρατου μέλου, τα συμφέροντα των πιστωτών, των πελατών και αυτό με φέρνει στο ζήτημα των τεχνητών διευθετήσεων, που είναι ε, ένα πολύ μεγάλο θέμα εάν δούμε την υπόθεση Μπόρμπιτ, ε, όπου το, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας λέει ότι μπορείτε να κάνετε εν τέλει ό,τι θέλετε ως επιχείρηση. Και τώρα η πρόταση της Επιτροπής βάζει κάποιους κανόνες, οργανώνει τη διαδικασία. Γιατί, για παράδειγμα, δεν ε, επιτρεπόταν σε όλα τα κράτη-μέλη να μεταβάλει την έδρα της μια επιχείρηση. Υπήρχαν κράτη-μέλη που δεν είχαν σχετική νομοθεσία. Αισθάνομαι ότι επαναλαμβάνω και πράγματα που ήδη ελέγχθησαν. Έρχομαι λοιπόν στο ζήτημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, που είναι στην καρδιά αυτής της οδηγίας. Προβλέπετε μια ειδική έκθεση να υποβάλλεται σε σχέση με την κατάσταση των εργαζομένων οι μέτοχοι, θα, υπό αυτή την έννοια δηλαδή οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοι ε, έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας. Θα υπάρχει μια ξεχωριστή έκθεση για τους εργαζόμενους, μια ξεχωριστή έκθεση για τους μετόχους. Επίσης έχουμε πολύ καλές διαδικα... Ε, προτάσεις για διαδικασίες για να... την καταπολέμηση τη απάτη. Αν προσπαθήσει κανείς να αλλάξει την έδρα του για να αποφύγει μια δίωξη, θα τον πιάσουμε. επίση, σε περίπτωση που μια επιχείρηση θέλει να μεταβάλει την έδρα τη και υπάρχει αντίδραση από την πλευρά των εργαζομένων, αυτό μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να παρέμβουν, έτσι ώστε τελικά να μην μπορεί να κάνει κανείς τη μετακίνηση για να παρακάμψει και να υποβαθμίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Κατά την άποψή μου αυτό είναι πολύ ψηλό επίπεδο προστασίας των εργαζομένων. Εγώ θα έλεγα ότι ε, επιχειρήσεις σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, οι άλλες χώρες που έχουν ε, υψηλή συμμετοχή των εργαζομένων δεν θα έχουν λόγο να κάνουν μεταβολή, να μεταφερθούν. Η προστασία των ε, δικαιωμάτων των μετόχων επίσης είναι υψηλή σε περίπτωση ψηφοφοριών εάν μια επιχείρηση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια χώρα που έχει υψηλή επίπεδο προστασίας ε, των μετόχων της μειοψηφία, δεν θα μπορέσει να μετακινήσει, να μεταβάλει την έδρα της για να το αποφύγει αυτό και να πάει σε μια άλλη χώρα με χαμηλότερο επίπεδο προστασίας. Και αυτό κατά την άποψή μου είναι σημαντικό στοιχείο της πρότασης. Θα έλεγα λοιπόν ότι η προστασία αυτή, σε αυτή την πρόταση είναι ουσιαστική και είναι και κάτι καινοτόμο. Δεν θα, προ... δεν θα προλάβει όλα τα προβλήματα. Επίσης, για το ζήτημα των εταιριών γραμματοθυρίδας, τις ψεύτικες εταιρείε που είναι ένα στοιχείο το οποίο βεβαίως ασκείται κριτική για αυτό από τις επιχειρήσεις. Αλλά κατά την άποψή μου το γεγονό ότι όλοι ασκούν κριτική για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη δείχνει ότι έχουμε καταλήξει σε καλό συμβιβασμό. Ε, γιατί όλοι είναι ικανοποιημένοι με κάποια στοιχεία και κάνουν κριτική σε κάποια άλλα. Άρα καλά πάμε. Συμφωνώ εν μέρη με την Business Europe ότι οι διαδικασίες για τους ελέγχους αυτούς θα μπορούσαν κάπως να περιγραφούν καλύτερα γιατί πράγματι πρέπει να προστατεύσουμε την ελευθερία της κίνησης του κεφαλαίου και της εργασίας που έχουμε και στις συνθήκες, ε, γιατί φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ε, μια καταρχήν υποψία έναντι της επιχείρησης που θέλει να μετακινηθεί. Επομένως, όπως είπε και ο συναδελφός μου, πρέπει να έχουμε ένα κοινό επίπεδο προστασίας σε όλες τις ε, σχετικές οδηγίες. Συμπερασματικά, έχουμε εδώ τις πιο σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει πάρει αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ε, έχουμε σε αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου και είναι η τελευταία ευκαιρία να ε, φροντίσουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί για μια μεγάλη επιχείρηση είναι εύκολο να μετακινηθεί. Ε, το ζήτημα είναι οι μικρές. Βεβαίως σε οποιοδήποτε νομοθετικό κείμενο μπορούν να γίνουν βελτιώσει, αλλά δεν πρέπει κανεί να ξεχνάει ότι καταλήγουμε σε ένα κείμενο μετά από συμβιβασμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε ε, δύο λεπτά για ερωταπαντήσει. Να ρωτήσω τον κύριο Κοβάσκε κατά πόσο θα ήθελα να μας αναφέρει την πηγή. Ναι, ευχαριστώ. Ρώτησα κάποιου αδέλφους για κάποιους υπολογισμού, ο καθηγητής Siegfried Holtz από το Επιστημονικό Κέντρο στο Βερολίνο που είπε ότι στην μελέτη, τελική μελέτη για την νομοθεσία που αφορά τις επιχειρήσεις θα βρείτε τα στοιχεία 499.000 αν δεν κάνω λάθος αναφέρει αυτή η μελέτη ευχαριστώ πάρα πολύ η κυρία Νίμπλερ έχει μια ερώτηση Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να αξιοποιήσω την ευκαιρία πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφου μα, τους εμπειρογνώμονε. Και η πρόταση αυτή πρέπει κυρίως, όχι μόνο αλλά κυρίως, να αποφευχθεί ο αθέμητος ε, φορολογικός ανταγωνισμός. γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να τροποποιηθεί το ε, φορολογικό δίκαιο γιατί χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο. Οπότε μέσω του εταιρικού δικαίου προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτές τις αθέμητες φορολογικές πρακτικές. Ρωτάω λοιπόν, θεωρείτε ότι οι προτάσεις της Κομισιόν, οι αλλαγές που μπορούμε να επιφέρουμε σε αυτές επιπλέον εμείς ως Κοινοβούλιο, ότι όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερο ισότιμο φορολογικό ανταγωνισμό, να αποφευθεί αυτό το forum shopping και να μην προσπαθούν τα κράτη να προσελκύσουν ε, με φορολογικά κίνητρα εταιρείε. Θεωρείτε ότι κάνουμε ένα έβημα προ τα μπρο με αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Ρέγνερ, σύντομα παρακαλώ. Στον κύριο Μόρο. Είπατε ότι πρέπει να τροποποιήσουμε το, την ιδεολογική σκέψη 7, ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καθορίζουν ποιε είναι οι πραγματικέ οικονομικέ δραστηριότητε. Μα δεν τα μεταφέρουμε όλα λοιπόν στα κράτη. Γιατί θα έχουμε 28 διαφορετικού ορισμού. Θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Απλώ έχει μεταφερθεί η νομική του θέση. Αυτέ ήταν οι ερωτήσεις. Θέλετε να απαντήσετε Ναι, για την πρώτη ερώτηση, κατάχρηση για τα φορολογικά. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πακέτο. Δεν μπορούμε με ένα σμπάρο να έχουμε δύο τριγώνια. Θα είναι κάπως δύσκολο. Πώς είναι η πρώτη φορά που λέμε ένα τέτοιο πακέτο για εταιρικό δίκαιο, το οποίο απευθύνεται και αφορά κατευθείαν τις φορολογικές καταχρήσεις. Βεβαίως πρέπει να δείτε προς τα που θέλετε να πάτε. Αν θέλετε να αποφύγετε τις φορολογικές καταχρήσεις, είναι περισσότερο έλεγχος από τις χώρες μέλη. Αυτό δεν είναι βέβαια τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον στέλνει ένα μήνυμα. Δεν ξέρετε ποτέ, τέλος πάντων, τι θα ορίσει κάθε χώρα μέλος ως αυτές τις ε, τεχνητές θα πρέπει λοιπόν να ψηλώσουμε τον πύχη. Και δεν είναι πανάκι, αλλά τέλος πάντων αποτελεί ήδη ένα μεγάλο βήμα μπροστά για αυτά, σε σχέση με αυτά που είχαμε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εδώ και 40 χρόνια, οπότε είναι ισχυρό μήνυμα. Παρακαλώ κυρία μου. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για τα δύο σημεία Όπως είπε ο συνάδελφος, δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα με αυτό το πακέτο. Πάντως, το αθέμητο φορολογικό πλεονέκτημα το αντιμετωπίζουμε και για το θέμα το φορολογικό ε, με ενσυχεί κάπως αυτός ο ορισμός του αθέμητου φορολογικού πλεονεκτήματος. Αυτό το αθέμητο αφήνει ακόμα πολλά ανοιχτά ζητήματα, ακόμα και για το ίδιο το φορολογικό ε, πλεονέκτημα, τι σημαίνει. Και αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να το συζητήσουμε για το ερώτημα της κυρίας Ρέγνερ για τις επιχειρήσεις γραμματοκιβώτιο. Σημαντικό αυτό, αλλά πρέπει να δούμε την ασυνέπεια μεταξύ αυτού του πακέτου και του θέματος των εταιριών αυτών. Πάντως, η ελευθερία εγκατάστασης προστατεύει τις επιχειρήσεις για την επιχειρηματική τους ε, δραστηριότητα σε όλες τις χώρες μέλη. και τι εξισώνει σε σχέση με τι άλλε επιχείρησει που είναι ήδη εγκαταστημένε στα πλαίσια αυτού του πακέτου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώ πρέπει να προχωρήσουμε στο τρίτο τμήμα που αφορά την ψηφιοποίηση και την προοπτική των επαγγελματιών της νομοθεσίας. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Λουκ ε, Χέντριξ Διευθυντή Επιχειρηματική Πολιτική και Εξωτερικών Σχέσεων στο UEAPME, e, η οποία κράθηκε οργάνωση εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε σήμερα. Όπως είπατε κι εσείς, είμαστε μια οργάνωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ένας κοινωνικός εταίρος για την ψηφιοποίηση και το πακέτο της στην πρόταση έχουμε εδώ τις ε, προσδοκίες των μικρομεσαίων δεν θα τις αντρέξουμε θα δείτε ότι το μόνο συμπέρασμα είναι η... το ότι τηρήθηκαν οι προσδοκίες μας με αυτή την πρόταση επίσης οι προτάσεις της ε, Κομισιόν συχνά τις επικρίνουμε, αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω είχαμε μια πολύ θετική διαδικασία διαβούλευσης και όλοι οι κοινωνικοί εταίροι που ήθελαν να σχολιάσουν είχαν δυνατότητα να το πράξουν. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στο αποτέλεσμα, γιατί νομίζω ότι το πακέτο της ψηφιοποίηση δεν είναι επίμαχο και νομίζω ότι έχει τη στήριξη όλων των εμπλεκομένων. Επιπλέον, ήταν απαραίτητο να τροποποιήσουμε το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο για την ψηφιοποίηση και θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε το ότι όλοι και οι μικρομεσαίες μπορούν να ωφεληθούν από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Τώρα για τα θέματα που απασχολούν τις μικρομεσαίες σε σχέση με την ψηφιοποίηση να πω καταρχάς ότι όταν μιλάμε για την ψηφιοποίηση. Αυτό αφορά κυρίως την απλούστευση. Απλούστευση όμως η οποία δεν θα πρέπει να είναι αυτός σκοπός. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία και νομίζω ότι και εδώ πέτυχε μια ισορροπία η Κομισιόν μεταξύ δηλαδή αφενός της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και της ε, καταπολέμησης της απάτης και διασφάλιση του θεμητού και αφετέρου της απεριόριστη οικονομική δραστηριότητα και της κάλυψης των αναγκών των επιχειρήσεων. Έχουμε λοιπόν εξασφαλίσει εδώ μια ισοτιμία. Πάντως παραμένει μια ανησυχία μας ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ελέγχων ταυτότητας και κλοπής ταυτότητας. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε πολύ υψηλέ προγραφές ευρωπαϊκές... για αυτούς τους ελέγχους που αφορούν την ταυτότητα. Και έχουμε και τους ελέγχους στο άρθρο 28 που περιλαμβάνουν τους ελέγχους στα υποκαταστήματα οι χώρε μέλη εδώ χαμηλώνουν τις προδιαγραφές τους και αυτό δεν είναι καλό. Επίσης στο 7 αναφέρουμε ότι ένα αντίγραφο ας πούμε του διαβατηρίου αρκεί και θεωρούμε ότι βεβαίως οπωσδήποτε δεν αποτελεί αυτό η υψηλή ευρωπαϊκή προδιαγραφή οπότε θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον την χρήση ηλεκτρονικής ε, ταυτότητας με το τσίπ δηλαδή. Επίσης πρέπει να υπάρχουν διαζώσεις έλεγχη, ταυτοπροσωπίας δηλαδή, και αυτό θα ήταν πολύ θετικό. Τώρα θα πάρω στα θετικά. Γιατί βλέπετε δεν έχουμε και τόσα αρνητικά σχόλια, τόσες επικρίσεις. Τα θετικά λοιπόν, που πιστεύω θα πρέπει να παραμείνω στην πρόταση, για πρώτη φορά εδώ μπορούμε να ε, συγκροτήσουμε επιχείρηση ηλεκτρονικά κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατόν. Αφετέρου όμω επιμένουμε για το γεγονό ότι αυτά τα συστήματα σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά. Γιατί βλέπουμε συχνά σε εθνικό επίπεδο όταν θεσπίζουμε λύσεις ηλεκτρονικές ότι τα συστήματα τα ίδια δεν μας επιτρέπουν να είμαστε αποτελεσματικοί και επίσης θα πρέπει να υπάρχει ένα help desk για τις μικρομεσαίες. Επίσης πολύ θετικό είναι το γεγονός ότι οι χώρες μέλη είναι υποχρεωμένες να παράσχουν υποχρεώσεις για την ενημέρωση και επίσης θα θέλαμε να τονίσουμε το ότι η παροχή νομικών συμβουλών πρέπει να αφορά και τους ε, συμβολεογράφους οι οποίοι βεβαίως θα είναι και ενημερωμένοι σωστά. Επίσης για το Μητρό των Επιχειρήσεων βλέπουμε ότι σε κάποιες ε, χώρες αυτό είναι απαγορευτικό παρόλα αυτά θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες, ώστε να έχουμε δηλαδή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα μας επιτρέπουν να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση στις ε, πληροφορίες. Και επ' αυτού καλωσορίζουμε το γεγονός ότι τα τέλη και τα κόστη θα πρέπει να είναι διαφανή θα πρέπει να είναι ορατά και να μην υπερβαίνουν το διοικητικό κόστος. Αυτό το αναφέρει ξεκάθαρα η πρόταση. Έχουμε όμω κάποιες ανησυχίες επειδή αναρωτιόμαστε πώς μπορεί κανείς να επαληθεύσει τη μη υπέρβαση διοικητικού κόστους γιατί αναφέρεται στο ψηφιακό βοήθημα ότι πρέπει να, έχουμε, να κάνουμε τα τωρινά διοικητικά κόστη. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή με την ψηφιοποίηση μάλιστα το κόστος ε, θα είναι χαμηλότερο από ό,τι πριν. Επίσης, πολύ θετική είναι η εφαρμογή της αρχής APAX. Εδώ στο εταιρικό δίκαιο το χαιρετίζουμε αυτό, αλλά ίσως να μην το ξέρετε. Εμείς εδώ και καιρό επιμέναμε για την εφαρμογή αυτής της αρχής από τις δημόσιες αρχές από 2005 κιόλα. Μπορώ λοιπόν να πω ότι είχαμε υπομονή και χαιρόμαστε που αυτή η αρχή της μιας φοράς, άπαξ, έχει ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πολύ θετικά λοιπόν, θαυμάσια πρόταση. Ίσως η Κομισιόν να έχει να έπρεπε να είχε πάει λίγο παραπέρα σε σχέση με την ψηφιοποίηση του εταιρικού δικαίου, αλλά τέλος πάντων φαντάζομαι ότι ταιριάζει και στην πολιτική και της Κομισιόν αλλά και των χωρομελών για την ψηφιοποίηση, γιατί εδώ στην ουσία δημιουργούμε ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον και είναι εξίσου σημαντικό οι χώρες μέλη να είναι σε θέση να διατηρήσουν τις νομικές τους παραδόσεις. Ταυτόχρονα ελπίζω ότι η σχέση αυτή μεταξύ των δύο ε, προτάσεων θα είναι ορατή, γιατί αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ σημαντική για μας για τις μικρομεσαίες και ελπίζω πάρα πολύ σύντομα να περάσει αυτή η πρόταση για ψηφοποίηση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από το τέλος της ε, θητείας, δηλαδή ώστε να έχουμε κάτι στο οποίο θα προσδοκάμε. Αυτά από μένα και ευχαριστώ. Θα έχετε και το έγγραφο με τις θέσεις μας τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ. Ο δόκτωρ Μάριους Κόλλερ τώρα, που είναι από το Συμβούλιο των Συμβολιογράφων της Ένωσης. Παρακαλώ 7 λεπτά. Ε, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη μου τιμή αλλά και χαρά που μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσω για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιοποίηση στο εταιρικό δίκαιο από πλευρά των Ευρωπαίων Συμβολιογράφων. Και συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές γιατί και εγώ θεωρώ ότι γενικά είναι θετική η στάση μου προς την πρόταση. Όπως ξέρετε και όπως λέει και το κείμενο της πρότασης σε πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης. Οι συμβολογράφοι παίζουν ρόλο κλειδί στη διασφάλιση και νομικής βεβαιότητας και για την αποφυγή καταχρήσεων καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής των εταιριών. Λοιπόν, τι ακριβώς κάνουμε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των επιχειρήσεων, του κύκλου ζωής. Επειδή είναι δημόσιο το λειτουργήμά μας, έχουμε το, το ρόλο να ελέγχουμε τα καταστατικά και ελέγχουμε και στέλνουμε μέσα στα πλαίσια των διαθρωμένων ηλεκτρονικών στοιχείων στέλνουμε στοιχεία στα επαγγελματικά μητρώα και δίνουμε πληροφορίες και στις ε, φορολογικές αρχές. Αν υπάρχει λοιπόν ε, ενδεχόμενο παράνομης δραστηριότητας ή απάτης, ξέπλυμα ο συμβολιογράφος φυσικά θα αρνηθεί να δράσει και θα ενημερώσει και τις ε, αρμόδιες ε, διοκτικές αρχές. Με την εξαίρεση της ίδιας της συμβολογραφικής πράξης, όλα τα άλλα βήματα γίνονται πλήρως ε, ψηφιπημένα στα κράτη-μέλη και αυτό αφορά και την επικοινωνία μεταξύ του συμβολογράφου και των δημοσίων αρχών όπως τα διάφορα δημόσια μητρώα. Αυτή είναι η διαδικασία προληπτικού ελέγχου ούτω ώστε οι εταιρείε να έχουν δημιουργηθεί σωστά, ούτω ώστε το καταστατικό του να είναι προσαρμοσμένο στι ανάγκε των ιδρυτών και ότι οι διαρθρωτικέ δομέ που θα γίνουν, ε, αλλαγέ που θα γίνουν κατά τη διάρκεια τη ζωή τη ε, επιχείρηση είναι επίση νομικά σωστέ. Περαιτέρω, οι πληροφορίε που στέλνει ο συμβολιογράφο στα δημόσια μητρώα και που μετά κοινοποιούνται στο κοινό είναι πλήρω αξιόπιστα και χαίρουν πλήρους εκτίμηση στα κράτη-μέλη για τις επιχειρήσεις και για τις ε, κυβερνητικές αρχές. Έτσι αποφεύγουμε χρονοβόρες ε, και ιδιαίτερα τα πανερές διαδικασίες για να δούμε ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος και ποιοι είναι οι νομικοί εκπρόσωποι μιας εταιρεία. Και παράλληλα, η χρήση εταιριών για παράνομους σκοπούς, όπως για παράδειγμα ε, ψευδή αυτοαπασχόλησης, ξέπλυμα χρήματος ή φόρο αποφυγή, τελικά παρεμποδίζονται αποτελεσματικά Ας εξετάσουμε τώρα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιο στενά. Από πιο κοντά δηλαδή. Αφήνει επαρκές περιθώριο η πρόταση στα κράτη-μέλη που έχουν ένα ε, καταξιωμένο τέτοιο σύστημα προληπτικού ελέγχου να μεταφέρουν αυτά τα συστήματα στην ψηφιακή εποχή. Γι' αυτό η πρόταση, κατά τη γνώμη μας, είναι εξαιρετική βάση για την περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση. Πιστεύουμε ότι βρήκε καλό τρόπο για να εφαρμόσει την ψηφιοποίηση στο εταιρικό δίκαιο χωρί να προκαλέσει δυσχέρειες στα κατεξιωμένα νομικά συστήματα των κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά, κατά τη γνώμη μα, κάποιε τροπολογίε ε, είναι αναγκαίε για να παραμείνουν αξιόπιστα τα επαγγελματικά μητρώα, τα μητρώα επιχειρήσεων και για να μην υπάρξει κατάχρηση των επιγραμμικών επιχειρήσεων. Και θα ασχοληθώ με τρία τέτοια θέματα. Πρώτον, Κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι σε όλη τη διάρκεια λειτουργία των επιχειρήσεων μπορούν να εμπλέκονται οι συμβολογράφοι. Οι επιγραμμικές διαδικασίες δεν θα πρέπει να ε, υπολείπονται των προδιαγραφών για την νομική βεβαιότητα και αξιοπιστία, ιδιαίτερα όσον αφορά διάφορες ε, προκαθορισμένε μορφέ εγγραφή. Η επιγραμμική ε, εγγραφή των επιχειρήσεων είναι υπερβολικά ευρεία μπορούν να συστήσουν εταιρείε ή άλλες εταιρείε, ε, καινούριε εταιρείε. Όσον αφορά το πρώτο θέμα, ότι οι συμβολογράφοι πρέπει να εμπλέκονται σε όλη τη λειτουργία των επιχειρήσεων, σε όλη του τη ζωή. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα λέει ότι οι συμβολογράφοι πρέπει να παρεμβαίνουν μόνο όταν συστήνεται μια εταιρεία. Η ανάγκη όμω για να δίδεται σωστή πληροφόρηση και έλεγχο αφορά ολόκληρη τη λειτουργία τη εταιρεία. Για παράδειγμα, όταν γίνονται αναδιαρθρώσει που πρέπει να μπουν στα Μητρώα. Για παράδειγμα, τροποποίηση του καταστατικού, μέτρα για το κεφάλαιο, συγχωνεύσεις ή και θηγατρικέ. Αλλιώ η και θηγατρικε αλλιως η ποιοτητα και η αξιοπιστία των ε, εταιρικών μητρών τίθεται εν κινδύνο. Κατά τη γνώμη μα, πρέπει να διευκρινιστεί στα άρθρα 13 και 28α και β ότι τα κράτη-μέλη έχουν κάθε δυνατότητα να κάνουν προληπτικούς ελέγχους νομιμότητας από τους ε, συμβολογράφους όταν γίνεται και η σύσταση της εταιρεία, αλλά και ε, η καταχώρηση υποκαταστημάτων. Και αυτό αφορά και την ε, δεύτερη ε, ρύθμιση για την διαμεθοριακή κινητικότητα των εταιριών. Οι υποχρεώσεις ενημέρωσης και τα προκαταρκτικά πιστοποιητικά για τις διασπάσεις. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό το άρθρο 13F λέει ότι ο έλεγχος νομιμότητας πρέπει να είναι μόνο εθελούσιος για το όνομα, το λόγο λειτουργίας και το καταστατικό. Το άρθρο 10 της οδηγίας του 2017 για το εταιρικό δίκαιο ε, προβλέπει υποχρεωτικό τέτοιο έλεγχο. Για να υπάρχουν ε, λοιπόν ε, αξιόπιστες εταιρικές συναλλαγές δεν θα πρέπει να υπολείπονται του κεκτημένου οι νέες αυτές ρυθμίσεις και επίσης και το, η προκαθορισμένη μορφή καταχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 13G λέει ότι ο προληπτικός έλεγχος που προβλέπει το άρθρο 10 θεωρείται ότι πληρούνται αν χρησιμοποιηθεί αυτή η προκαθορισμένη μορφή αλλά η προκαθορισμένη μορφή ε, σημαίνει πως δεν πρέπει να ελέγξουμε την ταυτότητα των ε, ιδρυτών σίγουρα όχι η νομιμότητα πρέπει να εξαρτάται και από ποιος είναι ο σκοπός. Δεν ε, μπορούμε λοιπόν να απαλείψουμε να απαλείψουμε την ε, ρύθμιση που υπάρχει στο προηγούμενο δίκαιο. Θα πρέπει να καταργηθεί λοιπόν η τελευταία πρόταση του άρθρου 13G παράγραφος 2. Νομίζω το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Τελευταίο. Ποδήλιο εφαρμογή της επιγραμμικής ε, σύστασης εταιριών το 13F είναι ιδιαίτερα ευρύ. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να την περιορίσουμε μόνο στην εγγραφή εταιριών από φυσικά πρόσωπα. Γιατί α δούμε τα σκάνδαλα LuxLeaks, ε, τα έγγραφα του Παναμά και τα έγγραφα του Παραδείσου. Αυτά έδειξαν ότι το επαγγελματικό μοντέλο των φορολογικών παραδείσων βασίζεται σε ε, μη διαφανείς εταιρείε που κρύβουν τους πραγματικούς ε, δικαιούχους. Γι' αυτό οι προτάσεις του FATF προτοποιούν κατά τέτοιων ε, διαδικασιών. Για αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι το να επιτρέπεται από άλλες εταιρείε ή από νομικά πρόσωπα να συστήνουν επιγραμμικά εταιρείε ε, είναι προβληματικό. Γιατί είναι δύσκολη η επαλήθευση εάν υπάρχουν αυτές οι άλλες εταιρείε και ποια είναι τα δικαιώματα των εκπροσώπων τους. Δεν είναι δυνατόν αυτά να γίνουν με ψηφιακά μέσα. Τέλος. Η δυνατότητα εξαίρεση ε, επιτρέπεται, μόνο για τι ανώνυμες εταιρείε, εξαίρεση από την επιγραμμική ε, καταγραφή. Αυτό θα πρέπει να επεκταθεί και σε ετερόρυθμες καταμετοχές, όπως για παράδειγμα οι, οι γερμανικές εταιρείες Commandit και by Action. Γιατί αυτές είναι τόσο περίπλοκες όσο και οι ανώνυμες. Δεν έχω άλλο χρόνο. Εμείς οι συμβολιογράφοι Είμαστε προετοιμασμένοι για περαιτέρω ψηφιοποίηση, αλλά για να επιτύχουμε αυτό το στόχο χρειάζονται κάποιε ασφαλιστικέ δικλείδε για να υπάρξει ταχύτητατη και αξιόπιστη καταγραφή των εταιριών στη σημερινή ψηφιακή εποχή προ όφελο όλων και των ε, μετόχων και των εργαζομένων και των πιστωτών και των δημοσίων αρχών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' από τον συνεισηγητή, τον εισηγητή μάλλον, για το θέμα αυτό, τον κύριο Σβιεύκα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας, τους προσκεκλημένους μας, που μας έδωσαν πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. αν και σύντομε οι παρουσιάσει, ήταν πολύ ενδιαφέρουσε και μα δώσετε μια εικόνα των απόψεών σα σχέση με την πρόταση τη Επιτροπή. Έρχεται μια διαδικασία μπροστά μας στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί να έχουμε στενή επαφή, να συνεχίσουμε να ε, συζητούμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις μέσα για ορισμένες από αυτές τις διατάξεις. γιατί κατά την άποψή μου το σημαντικότερο ζητούμενο είναι να προσαρμόσουμε τη λειτουργία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο σήμερα, στη, στη σύγχρονη εποχή. Και όλο αυτό βέβαια διασφαλίζοντα ότι θα συνεχίσει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, θα συνεχίσουμε να μπορούμε να εμπιστευόμαστε αυτά τα συστήματα και θα μπορούμε να καταπολεμήσουμε το ξέπλυμα μαύρου χρήματο ή την φοροαποφυγή μέσω φορολογικών παραδείσων. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και τους Ευρωπαίους συμβολιογράφους. Γιατί είναι γνωστή η ε, εντιμότητά τους, η γνώση τους για το αντικείμενο και επίσης το γεγονός ότι κατέχουν ε, θέσεις με τις οποίες ε, προσέχουν το δημόσιο συμφέρον. Έχω ένα ερώτημα προς τον εκπρόσωπο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με θορύβησε αυτό που είπατε ότι εάν ακολουθήσουμε εγγραφή στο Μητρό των Επιχειρήσεων επιγραμμικά, αυτό θα υπονομεύσει, θα μειώσει το επίπεδο των προτύπων που έχουμε αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη. Όπως εγώ γνωρίζω τα πράγματα, δεν γίνεται αυτό ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν μπορεί να μειώσει το επίπεδο των προτύπων που υπάρχει στα εθνικά κράτη-μέλη. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε πιο συγκεκριμένα λοιπόν τι εννοείται. Αυτό το πρώτο ερώτημα δεν έχουμε χρόνο για όλα τα ερωτήματα που θα να σα θέσω. Έχω ένα ερώτημα λοιπόν και για του ε, συμβολιογράφου. Είπατε ότι γίνονται έλεγχοι όσον αφορά την νομιμότητα σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωή μια επιχείρηση. Και είπατε επίσης ότι ε, έχετε μια πρόταση θα πρέπει να περιορίσουμε λέτε, την επιγραμμική εγγραφή μόνο στα φυσικά πρόσωπα. Ε, σωστά το έχω καταλάβει ή προτείνετε και κάτι άλλο σχετικά. Ευχαριστούμε κυρία Χάουταλα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους ε, εμπειρογνώμονες για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους. Πιστεύω ότι ένα ενδιαφέρον στοιχείο της πρότασης αυτής είναι ότι θα έχουμε στη διάθεσή μας πληροφορίες με τρόπο διαφανή και ε, αξιόπιστο για όλες τις επιχειρήσεις που ε, δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Και για να συμβεί αυτό, εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζητούμε να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό μητρό επιχειρήσεων τυποποιημένο. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για, από αυτού. Και μιας και δεν μπορώ να θέσω το ερώτημα ευθέως στην Επιτροπή, θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς μπορείτε να το φανταστείτε, γιατί δεν έκανε τέτοια πρόταση η Επιτροπή. Στο δεύτερο πάνελ αναφέρθηκε την κυρία Μωρό και θα ήθελα να επανέλθω το ζήτημα των διευθυντών. Ε, καλωσορίζω τη δυνατότητα που δίνεται στα κράτη-μέλη να αρνηθούν ε, μια επιχείρηση να ορίσει ως διευθυντή της κάποιο πρόσωπο το οποίο δεν έχει το δικαίωμα αυτό σε άλλο, άλλη, ε, άλλο κράτος μέλος, σε άλλη χώρα. Όμως το ερώτημά μου είναι πώς θα το γνωρίζει αυτό το κράτος μέλος. Ε, γιατί δεν έχουμε ένα διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό μητρό. Τα εθνικά μητρώα ίσως έχουν τέτοιες πληροφορίες, όμως πώς θα διαθέτουμε αυτές τις πληροφορίες και πώς θα είναι επικυρωποιημένες και πώς θα είναι ε, σωστές. Ε, θα ήθελα να ακούσω και από τους προσώπους αυτού του πάνελ ποιες είναι οι απόψεις τους για το θέμα. Και τέλος, πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την οδηγία έτσι ώστε να σταματήσουμε την κατάχρηση τους ελεύθερης ε, σύσταση επιχείρηση σε οποιοδήποτε κράτο μέλο, η οποία συμβαίνει σε ορισμένε περιπτώσει ακριβώ για να αποφύγει κανείς την φορολόγηση. Να δώσω το λόγο στους ομιλητές μας για να απαντήσουν. Εγώ για το ερώτημα του συγητή. Στο άρθρο 28 της πρότασης για την εγγραφή των παραρτημάτων. Εδώ είναι μια πρόβλεψη η οποία θα υπονομεύσει προ ε, βλέψεις που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Αυτό μου το επεσήμανε μία από τις συνεργαζόμενες οργανώσεις μας στη Γερμανία. Δεν γνωρίζω πολύ αναλυτικά πώς λειτουργεί το σύστημα στη Γερμανία. Αν σας ενδιαφέρει μπορεί να το μπορώ να το ψάξω και να σας δώσω πάλι ε, πιο αναλυτικές πληροφορίες. Για την ερώτηση της Κυρια Χάτουλα δεν μπορώ να απαντήσω ε, για εκ μέρους της Επιτροπής. Προσπαθούμε μέσω της ψηφιοποίησης να καταπολεμήσουμε την απάτη. Μπορούμε να το πούμε απλά. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μέσω των εντύπων θα πρέπει να μπορεί να συμβεί και μέσω των ψηφιακών μέσων. Ε, μέχρι εκεί το βλέπω εγώ. Όμως θα πρέπει η ψηφιοποίηση να είναι ουσιαστική, να είναι πραγματική. Για να μην οδηγηθούμε ε, σε, στην αύξηση των ψευδών πληροφοριών που μπορεί να υπάρχουν στο σύστημα εξαιτία τη ψηφιοποίηση. Και πιστεύω ότι το εργαλείο για να το, για να το εξασφαλίσουμε αυτό είναι ο έλεγχο τη ταυτότητα. Κύριο Σκέλλερ. Η πρώτη ερώτηση στην οποία θα ήθελα να απαντήσω είναι ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές που θα ήθελαν οι συμβολεογράφοι. Όσον αφορά την επιγραμμική εγγραφή, το online registration, πιστεύουμε ότι δίνεται αυτή η δυνατότητα ε, υπερβολικά ευρέω σε πολλέ περιπτώσει. Δίνεται, για παράδειγμα, η δυνατότητα σε νομικά πρόσωπα να συστήσουν επιχείρηση, ε, ε, εταιρεία για να συμβαίνει αυτό, για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να ελέγξει κανεί το ιδιοκτησιακό καθεστώ του νομικού προσώπου που συστήνει την εταιρεία και αυτό δεν μπορεί να συμβεί αποτελεσματικά online. Γι' αυτό ζητούμε η online ε, σύσταση εταιρεών να επιτρέπεται μόνο από φυσικά πρόσωπα, όπως εξάλλου συμβαίνει στην Εσθονία, που είναι μια χώρα η οποία είναι στην πρώτη γραμμή της ψηφιοποίησης και της χρήσης της πληροφορικής σε αυτόν τον τομέα. Έχουν, περιορίσει λοιπόν την ε, σύσταση εταιριών από φυσικά πρόσωπα. Δεύτερο ζήτημα είναι η σύσταση εταιριών από αντιπροσώπους. Και εδώ πιστεύουμε ότι είναι επικίνδυνο αυτό. Με την πρόταση της Επιτροπής έχουμε ήδη τη δυνατότητα η σύσταση να γίνει online. Επομένως, γιατί να χρειάζεται επιπλέον η σύσταση να γίνει και από κάποιον αντιπρόσωπο. Κατά την άποψή μας, είναι καλύτερα λοιπόν να περιοριστεί η δυνατότητα ε, online σύστασης εταιρεία μόνο στα φυσικά πρόσωπα και αυτοπροσώπως. Για το δεύτερο ερώτημα για την καταπολέμηση της απάτης. Βεβαίως, ένα από τα καθήκοντά μας είναι η καταπολέμηση της απάτης και πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε τη ταυτότητα των συναλλασσομένων και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την πρόταση αυτή και στον αγώνα κατά, κατά του ξεπλήματος μαύρου χρήματο. Ευχαριστώ. Δυστυχώ δεν έχουμε άλλο χρόνο να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές μας που ήρθαν σήμερα και επίσης να ευχηθώ καλή τύχη και στους δύο εισηγητές για αυτά τα ζητήματα. Ολοκληρώσαμε και με αυτό το σημείο της ημέρης της διάταξης. Ωραία αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε με το αναβριθέν σημείο 10. Κύριε Κάφμα θέλατε το λόγο για την ψηφορία, έτσι. Θέλετε να μιλήσετε τώρα. Ναι, ναι. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω ένα διαδικαστικό σχετικά με τον 174.2 και 3 του κανονισμού για συμβιβαστικές τροπολογίες και την ψηφοφορία. Στο άρθρο 9 έχουμε δύο συμβιβαστικές, 6α και 6β και νομίζω στον κατάλογο της ψηφοφορίας έχουμε τη λάθος σειρά επειδή ο 174 κανόνας λέει ότι η τροπολογία η οποία έχει πολύ από το αρχικό κείμενο θα πρέπει να θεθεί σε ψηφορία πρώτα. Από ό,τι θυμάμαι, χθες είχαμε μια πολύ περίπλοκη ψηφοφορία για τα πραγματικά δικαιώματα, οπότε θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον κανόνα ότι οι εναλλακτικές τροπολογίες πρέπει να ψηφίζονται πρώτα. Οπότε αυτό δεν φαίνεται στο κατάλογο της ψηφοφορίας και θα ήθελα να μάθω το γιατί. Οπότε θα ήθελα να μου το εξηγήσετε διαφορετικά. Θα επιθυμούσαμε να αλλάξουμε την σειρά της ψηφοφορίας για τις συμβαστικές 6α και 6β. Ευχαριστώ. Well, I think the, the... Πρόεδρος, η σειρά είναι σωστή για να διευκολύνουμε την διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Και η άποψη του εισηγητή ίσως ποια είναι να μας πει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τους σκιώδεις ε, με τους οποίους συνεργάστηκα πολλές εβδομάδες, μήνες ολόκληρους. Εργαστήκαμε σκληρά για να επιτύχουμε συμβιβασμούς. Ήταν πραγματικά σκληρή έντονη εργασία και ευχαριστώ πραγματικά τους συναδέλφους γιατί νομίζω ότι τελικά καταλήξαμε σε καλό αποτελέσματα. Και να ευχαριστήσω και τη γραμματεία για την ε, βοήθεια που μου έδωσε. Νομίζω ότι είναι σωστή η σειρά των ψηφοφοριών όπως προβλέπετε, γιατί ετέθησαν και προθεσμίες και στάλει ο κατάλογος ψηφοφοριών σε όλους τους κοιόδης ε, με το αίτημα να μας προτείνουν τροπολογίες. Και τώρα μετά τη λήξη της προθεσμίας έχουμε αυτή την πρόταση των σοσιαλιστών. Εγώ νομίζω ότι η πρόταση που αποκλίνει ε, πολύ περισσότερο πρέπει να διατυπώνεται έτσι όπως είναι. Πρέπει να έχει τη σειρά που έχει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είμαι στα χέρια σας, κύριε Πρόεδρε. Εάν θέλετε να τηρήσετε τη σειρά ή όχι, εμένα δεν με ενδιαφέρει, το ίδιο είναι. Πρέπει να ψηφίσουμε και τα δύο. Τώρα, το θέμα δεν είναι το να επιμείνουμε. Εγώ νομίζω πάντως ότι είναι σωστή η σειρά. Αλλά τώρα να, δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα. Παρακαλώ αποφασίστε κύριε Πρόεδρε, μπορώ να δεχτώ και τις δύο λύσεις. Η κυρία Ρέντα. Ναι, στηρίζω το αίτημα των σοσιαλιστών. Ο, το άρθρο 174 είναι σαφέ. Και υπάρχει και μία λογική να ψηφίσουμε πρώτα αυτό που αποκλίνει περισσότερο. Γιατί αλλιώς Κάποιοι συνάδελφοι μπορεί να χρειαστεί να καταψηφίσουν κάτι γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει σε μια μεταγενέστερη ψηφοφορία. Αν θέλουμε λοιπόν να περάσει το κείμενο με την ευρύτερη δυνατή συνένεση, πρέπει πρώτα να ψηφίσουμε αυτό που αποκλίνει περισσότερο από την ε, επικρατούσα άποψη. Αυτή νομίζω είναι η λογική διαδικασία. Γι' αυτό να αλλάξουμε τη σειρά στον κατάλογο ψηφοφοριών. Well, uh, Ωραία. Αφού η συγγήτρια δεν έχει αντιρρήσεις για τις αλλαγές, μπορούμε να αποδεχτούμε το αίτημα. Δεν έχω και εγώ αντίρρηση. So we begin. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχετε όλοι τοποθετήσει τις κάρτες ηλεκτρονικής ψηφορίας. Θα προσπαθήσουμε με ναι, ακόπτε πρόεδρος. So you will not be voting, Mr. Velkin, right? Okay. Δεν θα ψηφίσετε, κύριε Βέλτα, ε? Έτσι, ωραία. Very well. So... Πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. 25. Υπέρ. Απορρίπτεται, αλλά ας ξεκινήσουμε τους ηλεκτρονικούς ελέγχους. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. 149 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 153-154 ομού υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ναι. Ας ελέγξουμε. 158. 158. Ναι, ναι. Sorry, my mistake. Rejected, but... Λάθος, λάθος δικό μου. Απορρίπτεται. Αλλά είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα από εδώ που τα βλέπω. 157 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 160 και έκον 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται έκον 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται έκον 30 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 161 υπέρ. Κατά Αποχές. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται, λέει ο πρόεδρος. Α. 164. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 162 και έκον 31 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλ 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 και έκον 32 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλη 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 και 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78, 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 και 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 23 υπέρ. 23 λέει ο πρόεδρο, αλλά κάνει λάθο γιατί είναι 26. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εκρίνεται. Διακόπτει ο πρόεδρος. Can maybe somebody close the door or... Μπορεί κάποιος να κλείσει την πόρτα σας παρακαλώ.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

Ja, apa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

Σα ευχαριστώ. Uh, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί επιζήσαντες, survivors, λέει ο πρόεδρος, μιας και είμαστε σε δύσκολη σύνθεση τώρα, να σας προτείνω να αναβάλουμε την ψηφοφορία, να ψηφίσουμε για την αναβολή της ψηφοφορίας. στην έκτατη συνεδρίαση στο Στρασβούργο όπου θα προσπαθήσουμε να κανονίσουμε για μία Δευτέρα απόγευμα. Έχουμε σχολεία από κάτω από την αίθουσα. Τρίτη, τρίτη το απόγευμα τότε, Πρόεδρε. Τρίτη, τρίτη τα απόγευμα. Όχι Δευτέρα απόγευμα Στρασβούργο, τρίτη απόγευμα. Θα δούμε, θα δούμε τι θα μας δώσει και η υπηρεσία που ασχολείται με τις αίθουσε. Δεν εξαρτάται από μας. Εγώ είπα Τετάρτη τότε. Τετάρτη, Τετάρτη τότε. Αντιπρόταση από κάτω. Ε, ε, Πρόεδρος, κοίτα, και πάλι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε, δεν περνά από το χέρι μας πότε θα μας δώσουν τέλο πάντων αυτό το σλότ και την αίθουσα. Η γραμματεία μας εδώ θα υποβάλει το αίτημα και θα μας πούνε. Yes, hopefully, hopefully. Yes. Uh, and we will, we will, uh, we will resume the... Θα συνεχίσουμε με την 181 τροπολογία της πληροφορίας. 180, ε, όχι συγγνώμη, <laughs> ποιος είναι υπέρ της αναβολής της πληροφορία. υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οπότε συνεχίζουμε με ένα άλλο σημείο της ημερήσιας, το 29. Ανταλλαγή απόψεων με την παρουσία του δικαστηρίου σχετικά με το σχέδιο τροποποιήσεων του πρωτοκόλου αριθμός 3 περί του οργανισμού του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα καταρχάς να δώσω το λόγο στο, δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Τίμο Βόλκεν. Θα περιμένω, Πρόεδρε, ευχαριστώ, θα περιμένω λιγάκι να καθίσουν όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το λόγο αλλά και το δικαστήριο για την παρουσία του. Δεν θα αργήσω γιατί έχουμε καθυστερήσει, να περάσω κατευθείαν στα τρία κύρια θέματα αυτού του φακέλου. Καταρχάς για την κατάσταση της ενημέρωσης που έχουμε ε, μέχρι τώρα. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες λοιπόν και ποια είναι τα κυρία ζητήματα αυτά για τα οποία πρέπει να συζητήσουμε για τον φάκελο αυτό το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην πρόταση του λέει ότι παρά το γεγονός ότι είπε η έκθεση του 2017 ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση του πρωτοκόλου υπαριθμών 3 μετά από μεγαλύτερη σκέψη άλλαξαν άποψη αποδέχονται την τροποποίηση του πρωτοκόλου αριθμό, αριθμό, αριθμό 3 οπότε εγώ αναρωτιέμαι ποιοι είναι οι λόγοι που μας οδήγησαν στο να σκεφτούμε ότι αυτές οι αλλαγές στο αρχικό τμήμα της έκθεσης είναι απαραίτητες. Γιατί νομίζω περί αυτού συζητάμε τώρα. Δεύτερη ερώτηση. Κατά την υποβολή της πρότασης έχουμε αλλαγές στις δικαιοδοσίες ε, έχουμε μια αναδιοργάνωση των δικαιοδοσιών σε σχέση με το ελεκτικό συνέδριο, με το δικαστήριο κλπ. Αυτό ενδεχομένω να έχει αντίκτυπο να επηρεάσει κάποια δικαστικά μέσα και διαδικασίες. Ίσως να χρειαστεί να θεσπίσουμε διαδικασίες για να δούμε ακριβώς ποιες είναι παραδεκτές διαδικασίες και ποιες όχι. Οπότε το ερώτημα μου και πάλι είναι τι επιπτώσεις οικονομικές ή άλλης φύσης υπάρχουν εδώ μετά από αυτή την αλλαγή στην, στην διαδικασία αυτή και ποια είναι και η επίπτωση όσον αφορά την διάρκεια των διαδικασιών. Ας πούμε, η διαδικασία παραβίασης νομίζω υπό τον τωρινό κανονισμό εξετάζονται από άλλα δικαστήρια από αυτά που προβλέπονται. Έχουμε δηλαδή στην αρχή ένα πρώτο δικαστήριο που αποφασίζει και μετά έχουμε και ένα ανώτατο δικαστήριο το οποίο τέλο πάντων ε, τελεσίδικη. Αλλά νομίζω ότι οι διαδικασίε αυτέ θα παραταθούν, θα διαρκέσουν περισσότερο. Γιατί υπάρχουν κάποιες κυρώσεις που προβλέπονται υπό τις συνθήκες, αλλά αυτές θα εξασθενήσουν αν οι διαδικασίες είναι μεγαλύτερες από αυτές που προβλέπουν οι συνθήκες. Οπότε θεωρώ ότι το ενδεχόμενο εδώ είναι ότι οι διαδικασίες θα κρατήσουν πολύ περισσότερο και θα επηρεάσουν ακριβώς την ίδια την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτά είναι τα κυρία ερωτήματά μου και τρία κυρία σημεία που θα να δείξω. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους του δικαστηρίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερος που κρατήσατε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη παρά την ε, άσκηση εκένωσης του κτηρίου που κάναμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας δώσω λίγο το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει έρθει αυτή η πρόταση γιατί αυτό θα απαντήσει και σε κάποια από τα ερωτήματα που έθεσε ο εισηγητή. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η πρόταση αυτή είναι αποτέλεσμα ε, μιας ε, συζήτησης ουσιαστικής ε, που έγινε και από τα δύο τμήματα του δικαστηρίου και το Γενικό Τμήμα και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και ε, με την ευκαιρία ε, έχουμε ε, παρόντες εκπροσώπους, προέδρους και των δύο τμήματων που είναι στη διάθεσή σας για Και σας το λέω αυτό για να πω ότι έχουμε κάνει μια πολύ ουσιαστική εξέταση έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη διαχείριση των υποθέσεων που υποβάλλονται στο δικαστήριο. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των υποθέσεων και πρέπει να κάνουμε μια την καλύτερη δυνατή διαχείριση των πόρων που έχει το όργανό μας. Ε, θα πρέπει να σας δώσω μια εικόνα α, της κατάστασης της τρέχουσας του Γενικού Τμήματος και του Δικαστηρίου. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά το Δικαστήριο. Αυτό καταφέρνει να κάνει μια καλή διαχείριση των υποθέσεων, να ε, τυρά, τηρεί τις προθεσμίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τα προδικαστικά ερωτήματα και όσον αφορά την έκδοση των αποφάσεων. Όμω διαπιστώνουμε ότι έχει αυξηθεί ο αριθμό των υποθέσεων που υποβάλλονται στο δικαστήριο. Ε, δεν έχει φτάσει ακόμα στο ριό του, αλλά αυξάνονται. Κοιτούσα χτε τα στατιστικά στοιχεία μέχρι τις 20 Ιουνίου. Από 1η Ιανουαρίου μέχρι 20 Ιουνίου έχει δεχτεί 430 υποθέσεις. Το 2015 ήταν 309 υποθέσεις. Μετά κάθε χρόνο αυξάνεται κατά περίπου 40 υποθέσεις, 346, 380, τώρα φτάνουμε στα 430, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε μια ε, αύξηση 80% τελικά, ε, συνολικά. Και αυτή, αυτή η αύξηση των ε, υποθέσεων που εξετάζονται από το δικαστήριο δεν πρέπει να λειτουργήσει εις βάρος της ποιότητας ούτε εις βάρος της ταχύτητας της απονομής δικαιοσύνης. Και επίσης πρέπει να επισημάνω ότι αυξάνεται και η πολυπλοκότητα των υποθέσεων και επίσης όλο και περισσότερο γίνονται επίγουσες οι υποθέσεις που πρέπει, πρέπει, επί των οποίων να αποφασίσει το, το δικαστήριο και πρέπει να συνεχίσει να είναι σε θέση να το κάνει αυτό. και στο δικαστήριο ε, ε, για τους, ε, της διοίκησης, τριμπιουνάλ, έχει αυξηθεί ο αριθμός. Κατά 33% η αιτήσια αύξηση για το δικαστήριο, 28% για το δικαστήριο δημόσιας διοίκησης. Όμως, το Γενικό Δικαστήριο. Αυτή τη στιγμή Το Γενικό Δικαστήριο έχει μια δυνατότητα που δεν έχει το δικαστήριο. Έχει 28 α, δικαστές. Και μετά το Brexit θα μειωθεί ο αριθμός και των δικαστών και των, του γενικού, των γενικών εισαγγελέων. Στο Γενικό Δικαστήριο, επειδή το επιτρέπει αυτό η συνθήκη, έχει υπάρξει μια σταδιακή αύξηση του αριθμού των δικαστών των ε, δικαστών του Πρωτοδικείου, του Γενικού Δικαστηρίου, ανά μέλο. μέλος. Ε, έτσι λοιπόν, ήδη βλέπουμε μια έτσι, βελτίωση της κατάστασης στο Γενικό Δικαστήριο εξαιτίας αυτής της ενίσχυσης του, του αριθμού. Και θα σας δώσω κάποια στοιχεία. Η μέση διάρκεια στο Γενικό Δικαστήριο για όλες τις υποθέσεις από το 2013 στο 2017 από 27 μήνες έχει μειωθεί στους 16 μήνες πριν την ε, μεταρρύθμιση ήμασταν στους 48 μήνες 46 μήνες ήταν για τις υποθέσεις ανταγωνισμού παλαιότερα και τώρα έχουμε φτάσει στους 21 το οποίο σημαίνει ότι με την ενίσχυση του αριθμού των δικαστών στο Γενικό Δικαστήριο και παρά το, τα δυσκολίες που ε, προκύπτουν από την μεταρρύθμιση, καταφέρνει το Γενικό Δικαστήριο να εξετάζει τις υποθέσεις ε, τις δικές του με ποιότητα και με την ψυχραιμία που πρέπει. Ε, τα περισσότερα, οι περισσότερες υποθέσεις εξετάζονται από πενταμελή τμήματα ε, πριν τη μεταρρύθμιση αυτό δεν γινόταν, ήμασταν σε τριμελή τμήματα. Τώρα εκατοντάδε υποθέσει εξετάζονται από πενταμελή τμήματα. Καταφέρει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίζει, να εξετάζει περισσότερες υποθέσεις στο Γενικό Δικαστήριο και να λειτουργεί αποτελεσματικά. Με αυτές τις ε, συνθήκες έπρεπε να δούμε ποιες ήταν οι δυνατότητες που μας δίνουν οι συνθήκες για να ανταποκριθούμε και στις απαιτήσει και στις, ε, σε αυτό που αναμένουν από εμάς τα εθνικά δικαστήρια. Και καταλήξαμε στα εξή. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τι διαδικασίε επί παραβάση, παρέμβαση και επίσης για τις ε, εφέσεις, την προσβολή υποθέσεων του γενικού Δικαστηρίου ενώπιον του Δικαστηρίου. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ε, διαδικασίας επί παραβάση, προβλέπεται από το 256 άρθρο παραγράφος 1 της συνθήκης η δυνατότητα ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις να εξετάζονται από το Γενικό Δικαστήριο. Και αυτό σας προτείνουμε εν μέρη ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις, όπου ουσιαστικά η Επιτροπή προσφεύγει κατά κράτους μέλους, να τις μεταφέρουμε στο Γενικό Δικαστήριο με την εξαίρεση των υποθέσεων εκείνων στις οποίες αυτό που καταγγέλλεται είναι παραβίαση των συνθήκων συνθήκη και τι συνθήκε για τη λειτουργία τη Ένωση, γιατί αυτό είναι θεμελιώδε. Με, αυτή την εξέταση, με αυτή την εξαίρεση, κατά τα άλλα, ε, θα μπορούν οι υποθέσει αυτέ επί να εξετάζονται από το Γενικό Δικαστήριο. Στη διαφορετική περίπτωση, αν μιλάμε για τι συνθήκε, θα μπορούν να ε, εξετάζονται από το Δικαστήριο. Μόνο. Επίσης, μια άλλη εξαίρεση, ο τίτλος 5 ε, που αναφέρεται στην ελευθερία ε, μετακίνησης, ε, στις τέσσερις ελευθερίες και εδώ δεν προβλέπουμε μεταφορά. Όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις επί θα εξετάζονται από το Γενικό Δικαστήριο. Εμείς θεωρούμε ότι το Γενικό Δικαστήριο ε, έχει πλήρως τη δυνατότητα να το ε, πράξει αυτό, να εξετάζει αυτές τις υποθέσεις, γιατί επίσης είναι και ένα δικαστήριο το οποίο έχει την σχετική εμπειρία να ε, εξετάζει άμεσα τις εθνικές προβλέψεις, την εθνική νομοθεσία δηλαδή. Επομένως δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την ποιότητα των της εξέτασης των υποθέσεων και των αποφάσεων. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο μας το θέτει ο εισηγητής και είναι λογικό. Μήπως αυτό οδηγήσει σε αύξηση του χρόνου που χρειάζεται για να τελεσιδικήσει μια διαδικασία επί παραβάση. Αυτό το έχει εξετάσει το Γενικό Δικαστήριο ενδεχόμενο. Πρέπει να ε, γνωρίζουμε ότι η διαδικασία επί παραβάση είναι μια προκαταρκτική, αν θέλετε, μάλλον αυτό που κρατάει περισσότερο στη διαδικασία επί παραβάση είναι το σκέλος το επικοινωνία της διοίκησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αιτιολογημένες γνώμες, οι απαντήσεις κτλ. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που σας έλεγα ότι το Γενικό Δικαστήριο έχει διαποδείξει την ικανότητά του να ε, διεκπεριώνει γρήγορα τις ε, υποθέσεις του. Τρίτον, υπάρχει δυνατότητα για πιο ταχύ ρυθμή. Ε, διαδικασία σε περίπτωση που θεωρεί ότι το δικαστήριο ότι πρέπει να αποφανθεί επί της ουσίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα παραπέμπεται η υπόφαση στο Γενικό Δικαστήριο. Α, κατά τα άλλα, υπάρχει το ζήτημα το δικονομικό, το διαδικαστικό για τα γραπτά υπομνήματα. Και αυτές οι προτάσεις που κάνουμε έχουν ως στόχο να γίνεται πιο ε, ταχύρυθμα, αν θέλετε, πιο γρήγορα η διεκπαιρέωση της διαδικασίας επί παραβάση. Και θέλω να προσθέσω και το εξή που είναι επίσης σημαντικό. Ξεκίνησα λέγοντάς σας ποιος είναι ο αριθμός των υποθέσεων που το Γενικό Δικαστήριο πρέπει να... να συγγνώμη, το, το δικαστήριο χρειάζεται να εξετάζει. πρέπει να αναλάβουμε δράση, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα παρατείνεται ο χρόνος που θα χρειάζεται για να τελεξιδικήσει μια διαδικασία επί παραβάση του φόρτου εργασίας. Και αν δεν κάνουμε κάτι θα καταλέξουμε σε, σε καθυστερήσεις. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο για τις διαδικασίες επί αλλά επίσης και για τα προδικαστικά ερωτήματα. που είναι αν θέλετε το πιο σημαντικό στοιχείο της, της λειτουργίας του δικαστηρίου γιατί εκεί γίνεται ο διάλογος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των Εθνικών Δικαστών οι οποίοι σε συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ζητούν τη γνωμοδότηση του, του Δικαστηρίου του Ευρωπαϊκού. Και έτσι απαντώ και σε ένα άλλο ερώτημα του εισηγητή, τον Δεκέμβριο του 2017 είχε λεχθεί ότι δεν ήταν σωστό, ε, δεν χρειαζόταν να τροποποιηθεί ο οργανισμός. Όμως είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο να μπορεί το δικαστήριο να παραπέμπει στο γενικό δικαστήριο τα προδικαστικά ερωτήματα. Και ακριβώς αυτό ε, θεωρήθηκε ότι δεν πρέπει να, να, να γίνεται. Ε, είναι, πρόκειται για το 3 τέταρτα των υποθέσεων που εξετάζουμε. Είναι ουσιαστικό για την λειτουργία τη σωστή, και την σωστή εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και είχε ε, λεφθεί ότι η πιθανότητα να διασπαστεί αυτό σε δύο διαφορετικές, ε, διαφορετικά δικαστήρια να δημιουργήσει προβλήματα στην ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου. Και εν πάση περιπτώσει είχε κρίνει έτσι και η Επιτροπή και το Δικαστήριο. Η πρόταση όμως που κάνει τώρα το Δικαστήριο είναι πλήρως συμβατή με τα λεμιφθέντα το Δεκέμβριο του 2017 γιατί αυτό που προτείνουμε να μεταφερθεί στο Γενικό Δικαστήριο είναι οι υπόλοιπε υποθέσεις, δηλαδή η διαδικασία επιπαραλήψη ενώ οι υπόλοιπε παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο της πρότασής μας είναι ε, η δημιουργία ενός συστήματος υποθέσεων που διαπιστώνουμε ότι αυτή τη στιγμή αυξάνονται σε αριθμό, αν δούμε τις αποφάσεις τον αριθμό των σχετικών αποφάσεων στο δικαστήριο, τις περιπτώσεις των εφέσεων λοιπόν. Όπου και ιδιαίτερα όσον αφορά ζητήματα εμπορικών σημάτων. Δηλαδή, υποθέσεις τις οποίες μια διοικητική αρχή ανεξάρτητη έχει λάβει μια απόφαση η οποία προσβάλλεται και ε, στο, στο Γενικό Δικαστήριο. Και εδώ έχουμε συχνά προσφυγές ε, οι οποίες ε, καταλήγουν σε απόφαση πριν εκδώσει την απόφαση του του Γενικού Δικαστήριου. Ιδιαίτερα, για παράδειγμα, για το Ευρωπαϊκό Γραφείο για τα Εμπορικά Σήματα ή τον Ευρωπαϊκό ε, ε, ε, τέτοιου τύπου ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Σε αυτή τις περιπτώσεις λοιπόν το δικαστήριο επεμβαίνει για τρίτη φορά στην υπόθεση. Και η εμπειρία έχει δείξει ότι στις περισσότερες αυτές τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα της έφεσης είναι μια απόφαση όπου βασικά το δικαστήριο θεωρεί απαράδεκτη την προσφυγή. Και αυτό δεν είναι, δεν είναι καλή διαχείριση των χρήση των πόρων του δικαστηρίου. Για αυτές λοιπόν τις προσφυγές ζητούμε να δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερο σύστημα που θα εξετάζει το παραδεκτό τους. Για να εκθετηθούν τα επιχειρήματα από τον προσφεύγοντα, γιατί θεωρεί ότι την υπόθεση αυτή πρέπει να την εξετάσει το δικαστήριο. αν γίνουν δεκτές αυτές οι προτάσεις από το Συμβούλιο θα επιτρέψουν στο δικαστήριο να συνεχίσει να εστιάζει στα θέματα που πραγματικά αξίζουν τον κόπο. Ιδιαίτερα τα προδικαστικά θέματα όπου υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εθνικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που είναι στοιχείο κλειδί για τη σωστή λειτουργία του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτά Ελπίζω να μην ξέχασα τίποτα. Α, ναι. Ο εισηγητή στην αρχή της παρέμβασής του είπε ότι το Κοινοβούλιο περιμένει και άλλη πληροφόρηση. Νομίζω ότι θέλει και ένα δημοσιονομικό δελτίο. Γιατί αναφέρεται στις ε, δημοσιονομικές επιπτώσεις. Θα σας στείλουμε το δελτίο αυτό. Δεν νομίζουμε ότι θα έχει δημοσιονομική επίπτωση είναι απλώς ε, μεταφορά κάποιων υποθέσεων από το δικαστήριο στο γενικό. Άρα θα ε, κερδίσουμε και χρόνο όσον αφορά το παραδεκτό των ε, εφέσεων. Αλλά κυρίως θα είναι μια πολύ καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων του δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου. Θα σας στείλουμε λοιπόν, θα σας στείλουμε αυτό το δημοσιονομικό δελτίο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Ο κύριος Φως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Σνάλφος Ράντεφ, που είναι σκιώδης για το ΕΛΚ, δεν μπορεί να παρευρεθεί. Με παρακάλεσε να παρουσιάσω την άποψή του. Θα ήθελε περισσότερη πληροφόρηση και θα διαβάσω ότι μου έγραψε. Όσον αφορά τη μεταφορά προς το Γενικό Δικαστήριο για ορισμένες κατηγορίες ε, παραβάσεων, αυτό πρέπει να γίνεται με καλά περιγραφόμενες εξαιρέσεις που να βασίζονται στο 108, 258 και 259 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ένωσης. Το δικαστήριο, ωστόσο, θα έπρεπε να διατηρήσει την αρμοδιότητά του για τα θέματα που έχουν θεσμική και συνταγματική ισχύ. Θέλουμε λοιπόν ε, περισσότερες πληροφορίες. Ποιες ε, υποθέσεις μπορεί να έχουν ε, θεσμικές επιπτώσεις. Εκεί λέγεται ότι θα μπορούσε να αποφασίζει το δικαστήριο. Θα μπορούσε να το κάνει και αυτεπάγγελτα το, ειδικό, το Γενικό Δικαστήριο ή από το αίτημα, μετά από αίτημα εντός των διαδίκων, ενός των διαδίκων, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο όταν ε, ξεκινήσει η υπόθεση. Όπως και ο κύριος Ράντεφ, θεωρώ ότι μπορεί να έχουμε το ίδιο πρόβλημα όπως με τα προδικαστικά. Γιατί η ανάγκη για να αποφασιστεί ποιο θα το αντιμετωπίσει μπορεί να προκύψει αργότερα όταν θα καταστεί σαφής η πολυπλοκότητα του θέματος. Θεωρείτε ότι είναι δυνατόν να μεταφερθεί σε ένα μεταγενέστερο σχέδιο. Αυτό δεν θα παρατείνει την εξέταση της υπόθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο τον λόγο. Breton. Όχι, δεν έχω ρωτήσει. Ένα σχόλιο. Τα προδικαστικά θέματα είναι πολύ σημαντικά για τη λειτουργία του δικαστηρίου, γιατί περιμένουν τα εθνικά δικαστήρια. Πρέπει να εξετάζονται σύντομα. Πρέπει λοιπόν το δικαστήριο να διατηρήσει αυτήν την αρμοδιότητα. Θα αποφύγει διπλές εξετάσεις και νομίζω ότι θα καθησυχάσει και τους εθνικούς δικαστές να μπορούν να απευθυνθούν απευθεία στο δικαστήριο. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι για αυτή την ευκρίνηση. Για τα υπόλοιπα κατάλαβα ότι η μεγάλη καινοτομία που μας παρουσιάζεται είναι ένα σύστημα εξέτασης του παραδεκτού των ε, εφέσεων, ιδιαίτερα για θέματα εμπορικών σημάτων. Τέτοιες διαφορές ε, έχουν ήδη ε, εξεταστεί δυο φορές και οι περισσότερες τόσοι άλλως ε, απορρίπτονται. Νομίζω λοιπόν πως είναι μια καλή λύση. Ευχαριστώ πολύ. Το δικαστήριο θέλει να πει τίποτα. να απαντήσω στον κύριο Φως. Σύμφωνα με την πρότασή μας, το Γενικό Δικαστήριο σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας μπορεί να αποφασίσει να στείλει την υπόθεση στο δικαστήριο, όχι μόνο στην αρχή. Από τα κράτη-μέλη ζητάμε να το κάνουν στην αρχή, αλλά το Γενικό Δικαστήριο μπορεί να το αποφασίσει σε οποιαδήποτε φάση. Δεύτερον, Σα περιέγραψα την προηγούμενη διοικητική διαδικασία μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών, κράτου μέλου πριν το θέμα φτάσει στο, στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Θεωρούμε ότι όταν φτάνει στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, το κράτος μέλος ήδη ξέρει πολύ καλά το εύρο τη υπόθεση. Και είναι άριστα σε θέση να καταλάβει αν έχει έννοια να ζητήσει από το Γενικό Δικαστήριο να την παραπέμψει στο δικαστήριο. Υπάρχει λοιπόν ένα πρακτικό πρόβλημα. Και για τη διάρκεια της εξέτασης των υποθέσεων, σε τελευταία ανάλυση, θα ήταν πολύ καλύτερα να υιοθετήσουμε αυτή την μέθοδο. Γιατί αν ε, όλες τις υποθέσεις τις εξετάζει το δικαστήριο, τότε θα έχει φοβερό βάρος εργασία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Βέλκεν, εντάξει, σα ικανοποιεί. Η... Σας ικανοποιούν οι εξηγήσει. Ευχαριστώ για την ανταλλαγή απόψεων. Νομίζω ότι φώτισε κάπως την κατάσταση. Χαίρομαι που θα λάβουμε και το δημοσιονομικό δελτίο τι επιπτώσεις ενδεχομένως θα έχουν αυτές οι αλλαγές. Θα δω και τα επόμενα κείμενα που θα μου αποσταλούν, αλλά τέθηκαν και τα ερωτήματα του κυρίου Ράντεφ μέσω του κυρίου Φως, οπότε ίσως θα ήταν καλύτερα εμείς ως Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να σκεφτούμε μήπως θα ήταν καλύτερο να υπάρξει μια μελέτη αντικτύπου για να έχουμε πλήρη πληροφόρηση. Αυτό βέβαια θα είναι κάτι που θα το συζητήσω με τους κοιόδης. Αλλά μέχρι στιγμής ε, η ανταλλαγή βοήθησε και ευχαριστώ πολύ. Ωραία λέει ο πρόεδρος. Μήπως κάποιος άλλος επιθυμεί τον λόγο. Αν όχι, θα κλείσουμε το σημείο αυτό για σήμερα. Να σας ενημερώσω μόνο ότι οι επόμενες συνεδριάσεις θα γίνουν τη Δευτέρα 9 Ιουλίου από τις 3 μέχρι τις 6.30 και Τρίτη 10 Ιουλίου από τις 9 μέχρι τις 12.30. Ενδιάμεσα βέβαια θα έχουμε αυτή την έκτακτη συνεδρία στο Στρασβούργο για να συνεχίσουμε την ε, ψηφοφορία. Αναβάλουμε επίσης και τη συνάντηση των συντονιστών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους του δικαστηρίου που ήταν μαζί μας σήμερα.